Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε μπορούμε να αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Προσωρινά και ίσως όχι πολύ καλά θα αντικαταστήσω τον πρόεδρο Μπράινον Σίμψον που έχει καθυστερήσει λίγο εξαιτία των χιονοπτώσεων. Είναι, πάση περιπτώσει, ένα αεροπλάνο. Αλλά θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Εάν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις, θεωρώ ότι έχει εγκριθεί η μερίσια διάταξη. Τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, εάν δεν υπάρχουν ειδικέ παρατηρήσεις, θα θεωρήσω ότι έχουν εγκριθεί στο τέλος συνεδρίασης. Εξ ονόματός σας θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Φλουρέντζου, Υπουργό Επικοινωνίας και Δημοσίων Έργων της Απερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας, ο οποίος μετά το πέρας της Προεδρίας θα κάνει τον απολογισμό και ανταλλαγή απόψε με σας. Κύριε Υπουργέ, αφού παραγγείλουμε το καφεδάκι μας, μετά θα έχετε αμέσως το λόγο. Ε, έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, κύριε Αντιπρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω ενώπιον της Επιτροπής σας τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα των μεταφορών και παράλληλα να ακούσω τις δικές σας θέσεις και εκτιμήσεις. Η Κυπριακή Προεδρία κλήθηκε να διαχειριστεί και να προωθήσει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρωπαϊκές πολιτικές και επιδιώξεις που είναι άριχτα συνδεδεμένες με την ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Στον τομέα των μεταφορών, κατά το τελευταίο εξάμεινο, έτυχαν εξέτασης στο Συμβούλιο σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναμφίβολα στοχεύουν προς ένα πιο αηφόρο και αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών στην Ευρώπη στον τομέα των χερσαίων μεταφορών. Η Προεδρία εργάστηκε για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις συσκευές ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, ταχογράφη, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την καταπολέμηση της απάτης και την μείωση του διοικητικού άκθους. Το Συμβούλιο Μεταφορών του Οκτωβρίου ενέκρινε πολιτική συμφωνία επί της σχετικής πρότασης κανονισμού, ενώ οι συνεργάτες μου είχαν μια επικοδομητική συνεργασία με την εισηγήτρια της πρότασης, κυρία Τικάου, την οποία και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά. Είμαι βέβαιος ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο θα συνεχιστούν και θα ενταθούν επί Ιρλανδικής Προεδρίας με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Αναφορικά με την νομοθετική πρωτοβουλία για τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκινήτων, οχημάτων και των ρημουλκουμένων τους. Η Κυπριακή Προεδρία στη βάση της συζήτησης ανατολισμού που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών του Οκτωβρίου κατέληξε σε γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Πέρα από τις δύο αυτές νομοθετικές προτάσεις, δώσαμε έμφαση στην οδική ασφάλεια. Συγκεκριμένα, η Κύπρος φιλοξένησε στις 25 Ιουλίου του 2012 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τέταρτη Ευρωπαϊκή Μερίδα Οδικής Ασφάλειας η οποία με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας ήταν αφιερωμένη στους νέους. Η μερίδα κάτω από τη θεματική η ενεργός εμπλοκή των νέων στην οδική ασφάλεια είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση και δημιουργία κουλτούρας οδικής ασφάλειας ανάμεσα στους νέους. Δόθηκε έμφαση στην καλλιέργεια της κουλτούρας αυτής, διαμέσου της παιδείας και της εκπαίδευσης, καθώς και στη σημασία δημιουργίας κλίματος αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας ανάμεσα στην αστυνομία, και στους νέους ανθρώπους. Η εν λόγω ημερίδα αποτέλεσε μια σημαντική πλατφόρμα συζήτησης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και κυρίως ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους οι οποίοι ελοχεύουν από την ανεύθυνη οδήγηση. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που έχουν εξαχθεί από την ημερίδα αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τις εθνικές κυβερνήσεις καθώς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας ανάμεσα στους νέους τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, η Κυπριακή Προεδρία επικεντρώθηκε στην προώθηση της βελτίωσης των συνθήκων εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών για ένα πιο ασφαλές και υπεύθυνο εργατικό δυναμικό καθώς και σε μια πιο κοινωνικά υπεύθυνη ναυτιλιακή βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο Επικυπριακής Προεδρίας εξέτασε τις δύο νομοθετικές προτάσεις που άπτονται της μεταφοράς στην κοινοτική νομοθεσία των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας σε σχέση με τις υποχρεώσεις κρατών λιμένα και κρατών σημαίας που έχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί των συγκεκριμένων προτάσεων το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο Υπουργών του Οκτωβρίου. Εκτιμώ ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουν οι διεργασίες τόσο με τη δική σας Επιτροπή και ιδιαίτερα με τον Πρόεδρο Σίμψον ως εισηγητή της πρότασης για τις υποχρεώσεις του κράτους λιμένα όσο και με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και πιο συγκεκριμένα με την εισηγήτρια κυρία Μπέρες για επίτευξη συμφωνίας επί της Ιρλανδικής Προεδρίας. Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών η πλήρης εφαρμογή των λειτουργικών τμήματων εναερίου χώρου θεωρείται βασική συνιστόσα της διαδικασίας ολοκλήρωσης του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και ως εκ τούτου η Κυπριακή Προεδρία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο όλο θέμα. Στο πλαίσιο αυτό είχε συνδιοργανωθεί από την Κυπριακή Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάντηση υψηλού επίπεδου με τίτλο «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός. Ώρα για δράση» στη Λεμεσό στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2012. Η συνάντηση αποτέλεσε το φόρουμ για μια δυναμική συζήτηση αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση και την πρόοδο που θα έπρεπε να είχε σημειωθεί σε σχέση με τον έλεγχο του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Στη συνάντηση λοιπόν τόσο ο πρόεδρος Σίμψον όσο και άλλοι υψηλοί προσκεκλημένοι έστειλαν τα σωστά μηνύματα ως προς τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Ελπίζουμε ότι τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την ελόγω συνάντηση θα τύχουν της δέουσας προσοχής και σημασίας από όλους τους εμπλεκομένους προκειμένου να επιτευχθούν αυτά αποτελέσματα σε όλες τις συνιστώσεις του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού στο εγγύς μέλλον. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, το Συμβούλιο υιοθέτησε απόφαση σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ένωσης και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας που προβλέπει ένα γενικό πλαίσιο για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας Eurocontrol στο περιθώριο του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου υπογράφηκε η εν λόγω συμφωνία, η οποία αναμένεται ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο προσωπικά τον κύριο Σίμψον, όσο και την κυρία Φώστερ για την αγαστή συνεργασία που είχαν με τους συμβούλους μας εδώ στις Βρυξέλλες. Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών αερολιμένων είναι μια σημαντική πτυχή της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των αερομεταφορών. Η Κυπριακή Προεδρία επικεντρώθηκε στην εξέταση της νομοθετικής πρότασης σχετικά με τους κοινού κανόνες κατανομής των χρονοθυρίδων στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αποτελεί μέρος της νομοθετικής δέσμης για τους αερολιμένες. Επί της εν λόγω πρότασης, το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση τον Οκτώβριο. Έχω ενημερωθεί για την πρόσφατη ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο επί της δέσμης μέτρων μέσα από την οποία ανοίγει ο δρόμος για ουσιαστική διαπραγμάτευση και συμφωνία με το Συμβούλιο. Απευθύνω θερμές ευχαριστίες στους εισηγητές των τριών προτάσεων, κυρίους Ουγγίας, Λίχτεφριτ, Ενζασάτα για την αγαστή συνεργασία που είχαν με τους εκπροσώπους της Κυπριακής Προεδρίας. Επιπρόσθετα, στον τομέα των αερομεταφορών, η Προεδρία στη βάση σχετικής ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προώθησε σχετικά συμπεράσματα, τα οποία υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο σε σχέση με την εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εν λόγω συμπεράσματα αποτελούν τη βάση για συντονισμένη κοινοτική δράση στην προσπάθεια μετεξέλιξης του τομέα των αερομεταφορών σε διεθνές επίπεδο. Ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών προϋποθέτει σύγχρονες και αναπτυγμένες υποδομές. Η περαιτέρω ανάπτυξη και η σταδιακή ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων είναι ζωτική σημασίας για τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των αναγκών κινητικότητας των πολιτών και συμβάλλει στην ενίσχυση της δυνατότητας για ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δίκτυα αυτά μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την κοινωνική, εδαφική και οικονομική συνοχή μεταξύ όλων των περιφερειών της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό η Κυπριακή Προεδρία με βάση την μερική γενική προσέγγιση που είχε επιτευχθεί επιδανικής προεδρίας συνέχισε την εξέταση της νομοθετικής πρότασης για την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη Connecting Europe Facility ΣΕΦ επιτυχάνοντας σχετική πρόοδο. Η εξέταση της εν λόγω πρότασης έγινε στην νεοσύστατη ομάδα εργασίας φίλη της Προεδρίας η οποία δημιουργήθηκε με πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας για να διασφαλίσει τον οριζόντιο χαρακτήρα του περιεχομένου της πρότασης. Θερμές ευχαριστίες απευθύνω στον κύριο Ρικέ για τη συνεργασία που είχε με τους εκπροσώπους της Κυπριακής Προεδρίας. Η διαπραγμάτευση Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου για την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, καθώς και για τις τομεακές νομοθετικές προτάσεις, αναμένεται να συνεχιστούν επί Ιρλανδικής Προεδρίας. Ιδιαίτερα για την νομοθετική πρόταση που επιλαμβάνεται της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές κυρίους Κουμουτσάκο και κύριο Ερτούκ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαν με τους συνεργάτες μου. Πέρα από τη διαχείριση του πιο πάνω θεματολογίου, τολμήσαμε και θέσαμε προτεραιότητες, προωθώντας με επιτυχία πολιτικές που εκτιμώ ότι φέρουν πλέον το στίγμα της Κυπριακής Προεδρίας και που συμβάλλουν στην προώθηση της βιώσιμης και έξυπνης ανάπτυξης στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα έχουμε επιτύχει να επαναπροσδιορίσουμε την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από ειδική υπουργική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο οι Ευρωπαίοι Υπουργοί αρμόδιοι για θαλάσσια θέματα στην παρουσία του Προέδρου Μπαρόσο, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κυρίου Χριστόφια και της αρμόδιας Επιτρόπου Μαρίας Δαμανάκη διαμόρφωσαν και υιοθέτησαν τη διακήρυξη της Λεμεσού. Η διακήρυξη αυτή αναδεικνύει μια θαλάσσια και ναυτιλιακή ατζέντα για τη στήριξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η ατζέντα αυτή επικεντρώνεται σε υφιστάμενους αλλά και σε αναδυόμενους τομείς, στους οποίους υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για νέες θέσεις απασχόλησης και για ανάπτυξη. Πέραν αυτού, η διακήρυξη καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καλλιεργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορέσει να καμάσει η γαλάζια οικονομία. Τέλος, η διακήρυξη ζητά να αναπτυχθεί με γειτονικά τρίτα κράτη που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια λεκάνη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τομεακή και διατομεακή συνεργασία, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η προαγωγή διαλόγου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο εντός των νομικών πλαισίων που έχει θεσπίσει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η διακήρυξη της Λεμεσού αποτελεί ορόσημο για τον τρόπο που θα πρέπει να προωθήσουμε τις θαλάσσιες και ναυτιλιακές δραστηριότητες και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης, αξιοποιώντας πλήρως το θαλάσσιο πλούτο και τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης που απορρέουν από τις θάλασσες μας. Πρόκειται για μια αμυγός κυπριακή πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και των εκπροσώπων του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα τρία μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριο Κουμτσάκο, κυρία Λεπάς και κυρία Μάισνερ, που συμμετείχαν στη διάσκεψη και προσυπέγραψαν την επιτυχή έκφαση της διακήρυξης. Υπογραμμίζεται ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου ενέκρινε σχετικά συμπεράσματα μέσα από τα οποία υιοθετεί το περιεχόμενο της διακήρυξης. Τα εν λόγω συμπεράσματα αναγνωρίζουν ότι η διακήρυξη της Λεμεσού αποτελεί βασική συνιστόσα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που υποστηρίζει την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσα, μέσα από τη γαλάζια οικονομία. Επιπρόσθετα, επιδιώξαμε με επιτυχία τη σύζευξη δύο κεντρικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφιακού θεματολογίου και μεταφορών με την ανάδειξη του ρόλου της ψηφιακής τεχνολογίας στην αηφόρο ανάπτυξη των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν η πρώτη φορά που εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου οργάνωσε κοινή συνάντηση Υπουργών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο ρόλος των νέων και καινοτόμων τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός και κατέχει περίοπτη θέση στη Λευκή Βίβλο για την πολιτική μεταφορών. Μέσα από τα συμπαράσματα που υιοθέτησε η Κυπριακή Προεδρία και τα οποία χαιρετίστηκαν από το σύνολο των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητήθηκαν τρόποι που θα συμβάλλουν. Πρώτον, στην ελεύθερη χρήση πληροφοριών και δεδομένων ως βασικών στοιχείων στις ευφυείς μεταφορές. Και δεύτερον, στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών και την πολυτροπικότητα εντός και μεταξύ πόλεων υπογραμμίζεται ότι τα εν λόγω συμπεράσματα παρουσιάστηκαν από την Κυπριακή Προεδρία στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τα εφή Συστήματα Μεταφορών που φιλοξενήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην Αυστρία. Κύριε Αντιπρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, η Κυπριακή Προεδρία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για επίτευξη προόδου επί του ευρωπαϊκού θεματολογίου που κλήθηκε να διαχειριστεί. Επιπρόσθετα, οι πρωτοβουλίες που είχαν τεθεί από την Κυπριακή Προεδρία και αφορούσαν την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, καθώς και τους τονίστων των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, είχαν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να ευθυγραμμίζονται με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Εργαστήκαμε με συνέπεια, με τριοφροσύνη και πλήρη επίγνωση του ρόλου της προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έντιμου διαμεσολαβητή. Εργαστήκαμε με πλήρη σεβασμό στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι θεσμοί και οι αρχές της δημοκρατίας εκφράζονται κατά τρόπο υποδειγματικό. Μέσα από αυτή τη σημαντική εμπειρία της άσκησης της Προεδρίας, η Κύπρος απέκτησε εμπειρίες και περισσότερες γνώσεις στα ευρωπαϊκά δρόμενα που οπωσδήποτε θα αξιοποιηθούν. Επιβάλλεται να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με περισσότερο ζήλο και αποφασιστικότητα ως ενεργοί εταίροι συμβάλλοντας στον αδιαπραγμάτευτο στόχο για μια καλύτερη Ευρώπη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πλήρη και ειλικρινή συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στην Ιρλανδική Προεδρία και ιδιαίτερα στο φίλο μου Υπουργό Μεταφορών Λίο Βαράτκα ο οποίος ανέλαβε το πιδάλιο του Συμβουλίου από την 1η Ιανουαρίου του 2013. Παραμένω στην διάθεσή σας για να ακούσω τις δικές σας εκτιμήσεις και απόψεις και να απαντήσω στο μέτρο του δυνατού στα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστώ και για την υπομονή σας να με ακούσετε. Merci Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα δώσω το λόγο στους συντονιστές για ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ο κύριος Βέρνερ Κούν, ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την Κυπριακή Προεδρία και τον ε, Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Βλωρέντσου, για όλα τα θέματα που μιλήσατε. Έχουμε στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου μια ημερήσια διάταξη στην Επιτροπή μας. Ε, έχουμε ήδη κάποιες ε, πολιτικές αποφάσεις, στις οποίες όμως δεν έχει ακόμα υπάρξει Συνένεση. Αναφερθήκατε ε, για, την ενίσχυση του ενιαίου εναέριου χώρου και την ε, βελτίωση των, ε, του, των αέριων ελέγχων με τα FABs. Όμως τα κράτη-μέλη επιμένουν στην κατάστασή τους να έχουν δικές τους αρχές ε, εναέριου ελέγχου και ήταν απαραίτητο εσείς από την πλευρά σας ε, στην ε, Κυπριακή Προεδρία να πιέσετε και με τον Eurocontrol έγινε μια συμφωνία, υπογράφτηκε. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δέσμευσή σας. Επίσης να πω ότι ήταν πολύ θετικό το πακέτο roadworthiness, ειδικότερα στις τεχνικές, ε, στους τεχνικούς ελέγχους ε, για την ε, οδική ασφάλεια, τουλάχιστον από την πλευρά του Συμβουλίου, είχαμε μια κοινή θέση εδώ, την οποία στην Επιτροπή μας καταφέραμε να συζητήσουμε. Στο πακέτο για τα αεροδρόμια γνωρίζετε την κατάσταση. Έχουμε τις χρονοθυρίδες, Υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία για αυτό το θέμα. Η θέση του Συμβουλίου και η τριμερής ε, αυτή τη στιγμή για, τις, ε, για το ground handling επίσης ε, έχει οδηγήσει σε μια φάση που τώρα είμαστε και υπάρχει κάποια συμφωνία για τις υπηρεσίες εδάφους. Επίσης για τις θαλάσσιες μεταφορές που για την Κύπρο ως νησιωτικό κράτος και ναυτικό κράτος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο φυσικά. Θεωρώ ότι ε, είχατε πολύ θετική επιρροή. Επίσης, ε, οι συνθήκες διαβίωσης ε, και εργασίας στο, για τους ναυτικούς με βάση τη διεθνή τις υποχρεώσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και ειδικά για τις πατέντες που χρειάζονται, τα πιστοποιητικά που χρειάζονται στα πλοία για τις μηχανές, ε, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν, αλλά και για τον έλεγχο των κρατών σημαίας, ε, ε λιμένους, συγγνώμη. Τώρα το Συμβούλιο είναι αυτό που έχει την πρωτοβουλία. Έχουμε φυσικά και την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο, αλλά είναι σημαντικό αυτό το project σε επίπεδο επενδύσεων και υποδομών. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα ξεκάθαρο σήμα από το Συμβούλιο για το πώς αξιολογεί τις προτάσεις μας. Και ο κύριος Εκερός, ε, εισηγητής του Τσεφ, ε, στα οικονομικά ζητήματα ειδικά, ανέφερε ότι χρειαζόμαστε για τα επόμενα 7 χρόνια μια χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να γίνει η αρνητική κατάσταση, η οικονομική κατάσταση στα κράτη-μέλη μας θετική. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη τελικά να έχουν μια κοινή δημοσιονομική πολιτική ε, ώστε το 1% του προϋπολογισμού τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι τόσο πολύπλοκο. Αλλά θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες διαπραγματεύσεις των μεγάλων κρατών μελών. Η διακήρυξη της ε, Λεμεσού επίσης θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο, το αναφέρατε κιόλας. Είναι ε, μια, ένα στρατηγικό επίτευγμα στα πλαίσια της πολιτικής μεταφορών. Εξωτερικές μεταφορές επίσης είχαμε συγκεκριμένες αλλαγές. Ε, το μεσογειακό χώρο, να το αναφέρω, αλλά μάλλον δεν είναι αυτό στις δικές σας αρμοδιότητες κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι διαφορετικό κομμάτι εκεί προς αυτό το θέμα. Αυτά όμως παίζουν για την οικονομική ανάπτυξη πολύ σημαντικό ρόλο. Σας ευχαριστώ επίσης και για το θέμα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Ε, εργαστήκατε πολύ στεναρά και στο θέμα της, ε, των μεταφορών αλλά και στο θέμα του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για τη δέσμευσή σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ελκαντράουι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την εργασία που επιτελέστηκε και για την πολύ εμπεριστατωμένη ομιλία του σήμερα. Όντως, πέρασε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από όλα σχεδόν τα θέματα. Τους φακέλους που ολοκληρώθηκαν, κάποιου άλλους, τους ταχογράφους, ε, ε, και άλλα θέματα. Το θέμα της διευθέτησης των ταχογράφων είναι πολύ σημαντικό για την οδική ασφάλεια και νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο τις υπάρχουσες τεχνολογίες που μπορούν να μας βοηθήσουν. Και έτσι θα καταπολεμήσουμε και τις απάτες. Θα πρέπει όλοι να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Η Οδικές μεταφορές λοιπόν θα πρέπει να προσαρμοστούν στα σημερινά δεδομένα ώστε όσοι εργάζονται στον κλάδο αυτό να μπορούν να έχουν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτό όσον αφορά τους ταχογράφους. Τώρα, όσον αφορά την εναέρια κυκλοφορία και το σχετικό πακέτο Ακόμη έχουμε διάφορες ε, φακέλους για την ηχορύπανση, τις χρονοθυρίδες, άλλα διάφορα θέματα που μας απασχολούν και νομίζω ότι από την μεριά μας, από το Κοινοβούλιο, μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ένα λιγότερο θετικό νέο, το οποίο βεβαίως δεν έχει σχέση με την νομοθεσία την οποία εσείς εξετάζετε, είναι αυτό το οποίο αφορά την εφαρμογή των συμπεφωνημένων και κυρίως σκέφτομαι το κοινό εναέριο χώρο. Στις 5 ε, Δεκεμβρίου έπρεπε κάποιες αρχές να τεθούν σε ισχύ, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα απολύτως. Και όλα αυτά έχουν σχέση με την νομοθεσία που ήδη είχαμε υιοθετήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να είναι λοιπόν τα πράγματα σωστά θα πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι αρχές οι οποίες υιοθετούνται να εφαρμοστούν. Οι συμφωνίες θα πρέπει να γίνονται συμφαστές και το συμπέρασμα που μπορούμε να αποκομίσουμε είναι ότι όλοι μπορούν να επωφεληθούν από την σωστή εφαρμογή των κανόνων. Είναι λυπηρό που δεν χρησιμοποιούν ε, την υπάρχουσα νομοθεσία όλες οι χώρες, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του ΑΣΕΦ, καθώς επίσης και των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αντικειμενικοί όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών στην Ευρώπη. Πρέπει να προχωρήσουμε με τρόπο αντικειμενικό να καταλήξουμε τελικά σε μια αποτελεσματική, καλά, καλώς λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Και καταλαβαίνετε ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντικά ως προς αυτό. Μέχρι στιγμής έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και στηριζόμαστε και στη δική σας υποστήριξη τους επόμενους μήνες, στα πλαίσια της συμμετοχής σας στο Συμβούλιο δηλαδή, προκειμένου να μας βοηθήσετε, ιδίω όταν βλέπουμε την κατανομή του προπολογισμού, όπου ουσιαστικά αναφερόμαστε σε δισεκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια του προπολογισμού. Δεν θα ήταν λογικό να δαπανίσουμε πάρα πολύ χρόνο δημιουργώντα νέου κανόνε για τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, αν δεν έχουμε εξασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότηση. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχάς να έχουμε τον κατάλληλο προπολογισμό για τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και για τις ευρωπαϊκές υποδομές. Θα ήθελα επίση να επωφεληθώ τη ευκαιρία αυτή που μου δίνετε, προκειμένου να σα ευχαριστήσω για την εξαιρετική σα εργασία και προσβλέπουμε στην συνέχιση τη συνεργασία μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε Καντράουι. Εξ ονόματος των Φιλελευθέρων, ο κύριος Μπενέν έχει το ρόλο. Εκτός μικροφώνη παρέμβαση. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι έχουμε προχωρήσει στην ημερήσια διάταξη. Αναφερόμαστε στην έκθεση του κυρίου Καμάλ. Όχι, κοιτάξτε, αν δεν να κάνετε κάποια δήλωση ή κάποια παρατήρηση όσον αφορά την παρέμβαση του κύριου Υπουργού, τότε το λόγο θα τον πάρει κάποιος άλλος. Κύριε Μπενιόν, επ' αυτού θέλετε να μιλήσετε σχετικά με τη δήλωση του Υπουργού. Όχι, όχι. Δεν ήμουν προετοιμασμένο. Νόμιζα ότι είχαμε προχωρήσει στην ημερήσια διάταξη και ήμουν έτοιμο να μιλήσω για κάποιο άλλο σημείο. Συγγνώμη, δεν είχα ενημερωθεί. Σα το συγγνώμη. Εξ ονόματο των Πρασίνων, το λόγο έχει ο κύριο Κράμερ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την ε, Κυπριακή Προεδρία για την παρουσίασή της. Ε, όλα τα θέματα που αναφέρατε θα τα θίξω ε, σύντομα. Η συνάντηση στη Λεμεσό ήταν πολύ σημαντική, αλλά όπως υπόθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι επικεφαλής κρατών ε, και κυβερνήσεων αυτοί οι ίδιοι παραβιάζουν την νομοθεσία που ε, έχουν υιοθετήσει. Θα έπρεπε στις 5 Δεκεμβρίου να μπει η νομοθεσία σε ισχύ. Είναι μια ρύθμιση που ρυθμίζει τη μείωση των ε, εκπομπών, έχει να κάνει με την προστασία του κλίματος, όμως δεν γίνεται. Και αναρωτιέμαι τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Αυτοί που φτιάχνουν τους νόμους αδιαφορούν. Δεν μπορούν αυτοί οι ίδιοι να εφαρμόσουν αυτά που λένε. Πώς θα γίνει τότε συζήτηση, γιατί δεν το κάνουν αυτό που πρέπει έτσι απλώς. Εγώ είμαι από τη Γερμανία. Γιατί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της, Ομοσπονδιακής Γερμανίας δεν κάνει αυτό που έχει εκ των προτέρων. Ε, αποφασίσει και για το οποίο άσκησε πίεση να ληφθούν αποφάσεις έτσι ώστε να κερδίσουν όλοι τελικά. Δεν είμαστε μέλη των ε, ομάδων συζήτησης, δεν είναι διαφανείς αυτές οι ομάδες, αλλά πραγματικά τι σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Ο κάθε πολίτης στην Ευρώπη που ζει σε ένα κράτος ε, δικαίου πρέπει να ακολουθεί ε, τους νόμους, αλλά αυτό δεν ισχύει για τους ε, υψηλούς ας πούμε εκπροσώπους του Συμβουλίου. Ίσως μπορείτε να πείτε κάτι γι' αυτό. Τώρα για τις υπηρεσίες εδάφους, τις έχει, γίνει, έχει απορριφθεί με μεγάλη πλειοψηφία το θέμα αυτό και συζητούμε σήμερα στη μερίσια διάταξη αυτό το θέμα. Θεωρείτε λοιπόν, αν προστρέξω σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι οι υπηρεσίες εδάφους ε, που τώρα ε, στην ουσία έχουν να κάνουν με τρία αεροδρόμια ε, και θα είναι μια ρύθμιση που για πολλά χρόνια για τα ευρωπαϊκά κράτη Ίσως δηλαδή να μην είναι σωστό τελικά να ασχολούμαστε με τρία αεροδρόμια και να επηρεάζουμε όλα τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι είναι χάσιμο χρόνου. Η τρίτη παρατήρησή μου έχει να κάνει με τα περιφερειακά αεροδρόμια. Τη συζητήσαμε σε μια σχετική έκθεση και πήραμε κάποιες πληροφορίες ε, από το αεροδρόμιο του Κάσελ. Από το Κάσελ μπορεί κανείς απευθείας με το αεροδρόμιο να πάει ε, στο Φραγκφούρτη σε μία ώρα και 38 λεπτά και από εκεί μπορεί απευθείας να πάει σε πάρα πολλούς προορισμούς. Όμως ε, η κυβέρνηση του κυρίου Κόχ ε, στην περιφέρεια αυτή έφτιαξε και ένα περιφερειακό αεροδρόμιο κοντά στις Φραγκφούρτης και από εκεί φεύγουν κάθε εβδομάδα 12 αεροπλάνα, εκ των οποίων ε, τα περισσότερα είναι από την XL Airways, που είναι μια αφαιρέγγια εταιρεία. Επίσης στο Σάρμπρουκεν υπάρχει ένα τέτοιο περιφερειακό αεροδρόμιο. 400... Αυτό το αεροδρόμιο έχει ένα έλλειμμα 5,5 εκατομμύρια, τα οποία ε, πρέπει ε, να καλυφθούν με 120 εκατομμύρια ε, συνεισφορά από τους πολίτες. Θεωρείτε ότι αυτό ε, είναι σωστό, δεν είναι τα χρήματα το θέμα. Ποια είναι η αρχή που υπάρχει στην ε, Ευρώπη, το user pays principle, ο χρήστης πληρώνει. Όλοι οι στόχοι και οι αρχές πραγματικά παραβιάζονται. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, συζητείτε αυτό το θέμα στο Συμβούλιο, έχετε κάποια θέση γι' αυτό και ποια είναι τα επιχειρήματα που ακούμε. Ε, μπορεί να κάνουμε οικονομίες ε, στην παιδεία και σε άλλους τομείς, αλλά να δίνουμε χρήματα βέρτα για τα αεροδρόμια. Ε, είναι σωστό. Τώρα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, πριν από τα Χριστούγεννα υιοθετήσαμε μια, ένα και η ερώτησή μου σε εσά είναι ότι δεν, ότι δεν θεωρείτε ότι κάπου πρέπει να πούμε ότι έχουμε τόσα χρήματα, γιατί δεν ξέρουμε και πόσα είναι τα χρήματα, ίσως έχουν μειωθεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τα project που υπάρχουν ή θεωρείτε ότι το ευχολόγιο που σας ε, δώσαμε ε, είναι αυτό που πρέπει τελικά να γίνει. Γιατί τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχει γίνει ε, τίποτα. Επίσης ε, για τους σιδηροδρόμους έχουμε μια πρόχειρη δουλειά και αυτό είναι μια προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μάθω πώς συζητείτε το θέμα στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Στον κύριο Κόλιτσεκ τώρα θα στο λόγω μέρους της Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κυπριακή Προεδρία. Ξέρω ότι η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή διέρχεται μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και θα ήθελα να πω ότι η Κυπριακή Προεδρία παρόλα αυτά έκανε εξαιρετική δουλειά για όλα τα θέματα που αφορούν τις μεταφορές. Κυρίως το θέμα των ταχογράφων είναι πολύ σημαντικό και για τις ε, ε, μεταφορές εμπορευμάτων. Είναι πολύ σημαντικό για τους ε, οδηγούς των φορτηγών και κυρίως των μεγάλων φορτηγών. Η ασφάλεια επίσης είναι σημαντικό θέμα. Πολλές φορές εργάζονται σαν σκλάβοι 10 με 12 ώρες την ημέρα. Πολλές φορές ε, κοιμούνται μέσα στο φορτηγό του, στην άκρη του δρόμου. Οι συνθήκες λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολες και τα θέματα ε, όλα αυτά και η προστασία τους είναι πάρα πολύ μεγάλα. Κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τι ακριβώς γίνεται με τους οδηγούς των μεγάλων φορτηγών. Επίσης, το θέμα της κατάρτισής τους θα πρέπει να εναρμονιστεί, διότι νομίζω ότι τα περισσότερα δυστυχήματα και ατυχήματα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα της ασφάλειας και κατάρτισης των οδηγών. Όλοι οδηγούμε. Ε, αλλά αν κάποιος οδηγήσει ε, όπως ε, η επαγγελματίας οδηγεί των φορτηγών 80.000 χιλιόμετρα το δρόμο, ε, στο δρόμο ετησίως καταλαβαίνετε πόσο τυχεροί είναι όσοι δεν παθαίνουν κανένα τύχημα στο τέλος. Και ξέρω ότι έχει κάνει πολλά η δική σας προεδρία. Ίσως και η επόμενη. Δεν ξέρω όμως αν το θέμα αυτό σας ενδιαφέρει. Μιλούμε εδώ και χρόνια για τα έργα υποδομών και μέχρι τώρα δεν αν ότι έχει γίνει είναι επαρκές. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε λογικές λύσεις και να κάνουμε ό,τι μπορούμε κυρίως για να βελτιώσουμε την ασφάλεια και να ενοποιήσουμε την νομοθεσία. Τώρα, για τις εναερίες μεταφορές. Έχουμε κάνει πολλά για την ηχορύπανση, για τις χρονοθυλίγες. Δεν ξέρω όμως αν έχουμε κάνει σε θέματα ρύπανσης πολλά πράγματα, σε θέματα εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος. Πράγμα πολύ σημαντικό. Και γενικότερα αν έχουμε κάνει κάτι για να προστατεύσουμε το περιβάλλον από τη ρήπανση. Δεν νομίζω ότι έχουμε επιτελέσει μεγάλη πρόοδο. Ξέρω ότι κάποιες εταιρείες ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν μέτρα. Το θέμα των υπηρεσιών εδάφου επίσης είναι ένα θέμα που μας ε, απασχολεί. Ε, και εδώ προβλέπεται απελευθέρωση, όπως και στους λιμένες, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί ώστε να παρέχουμε την κατάλληλη προστασία στους εργαζόμενους για να μην στείλουμε αρνητικά μηνύματα. Όσον αφορά τα λειτουργικά μπλοκ, τα FABs. Ξέρω ότι ασχολούμαστε εδώ και 15 χρόνια με την ενοποίηση του εναερίου χώρου και οι συμφωνίες οι οποίες έχουν ε, ε, ήδη γίνει, δεν ξέρω πώς εφαρμόζονται. θύμω το θέμα της ε, εναερίου χώρου της κεντρικής Ευρώπης είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να λύσουμε και να καταλήξουμε σε συμφωνία. η κεντρική Ευρώπη ίσως είναι το πιο κρίσιμο μέρος αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω αν το όλο πράγμα θα μπορέσει να το επιλύσει επιτυχώς η Ιρλανδική Προεδρία. Εκτιμώ την πρωτοβουλία της ε, Λεμεσού για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές. Πρέπει να σας πω ότι και οι εσωτερικές ε, πλωτές μεταφορές ε, είναι πολύ σημαντικές ε, για χώρες όπως η δική μου. Ο Ρήνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις ε, πλωτές μεταφορές. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα κάνουμε κάτι στην Ευρώπη που θα είναι στον τομέα αυτό εποφελές για όλους. Οι πλωτές μεταφορές, όπως ξέρετε, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και στον τομέα αυτό δεν έχει ίσως δοθεί η κατάλληλη σημασία. Και ο Δούναβης, εκτός από το Ρήνο, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα των πλωτών μεταφορών μέσω του Δούναβη, τόσο μεγάλου ποταμού αυτού. Και και άλλων σημαντικών ποταμών στην Ευρώπη η Κυπριακή Προεδρία βεβαίως συνειδητοποιεί ότι οι μόνες σημαντικές μεταφορές δεν είναι οι θαλάσσιες και οι πλωτές είναι σημαντικές. Αυτό είναι σημαντικό. Σε όλους τους τομείς, σε βάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις. Επενδύσεις οι οποίες θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν πολύ Και βεβαίως τα κονδύλια που θα διαχειριστούμε θα πρέπει να τα διαχειριστούμε σωστά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες. Και αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σωστά, θα πρέπει να διαθέσει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για να μπορέσουμε να έχουμε αναθέρμανση της οικονομίας και ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και δεν θα πρέπει να το υποτιμήσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουν υπόψη οι μεγάλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κόλιτσεκ. Ο κύριος Κοχ και μετά ο Υπουργός. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την ε, πολύ καλή παρουσίαση όλων ε, των ε, συνεδρίων και των εκδηλώσεων που έχετε εκδηλώσει. Είδαμε τις είδαμε τις, τα αποτελέσματα. Είχαμε την υποχρέωση το 2015 να έχουμε ε, με ένα μεταβατικό διάστημα, όμως δεν θα τα καταφέρουμε γιατί για εμπορικούς λόγους τα κράτη-μέλη ε, το έχουν θάψει το θέμα της ασφάλειας. Επίσης, για τις ε, ψηφιακές τεχνολογίες υπάρχουν ας πούμε συστήματα που βοηθούν κάποιον που θα κοιμηθεί στο τιμόνι. Αυτό πραγματικά είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε εντατικά ε, και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τον κύριο Υπουργό, ο οποίος θα απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε θα προσπαθήσω να απαντήσω συνολικά τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις οι οποίες έχουν τεθεί έχοντας υπόψη και τον χρόνο ο οποίος είναι περιορισμένος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα καλά σας λόγια για το έργο που έχει παράξει η Κυπριακή Προεδρία και για την εκτίμηση που έχετε εκφράσει προς την εργασία την οποία έχουμε επιτελέσει ως Κυπριακή Προεδρία. τα μηνύματα μέσω της Συνόδου της Λεμεσού τον Οκτώβριο έχουν δοθεί, θα έλεγα μάλιστα έντονα, τόσο από τον κύριο Σίψον όσο και από τον κύριο Γκάλας. Εξαρτάται τώρα από εμάς, τα κράτη-μέλη, να υλοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Στο συνέδριο της Λεμεσού έγινε αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και συζητήθηκαν στην παρουσία του κυρίου Σίμψον και του κυρίου Κάλλας αλλά και του συντονιστή για τα ΦΑΠΣ οι μελλοντικές ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Επίσης όσον αφορά και πάλι στις παρατηρήσεις του κ. Κράμερ για τα ΦΑΠΣ, πρέπει να είμαστε συνεπείς με τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις και πρέπει να εργαστούμε σκληρά για την παρακολούθηση και εφαρμογή του κοινοτικού και Ιδιαίτερα σήμερα που διερχόμαστε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Όσον αφορά το αεροπορικό πακέτου. Έγινε σημαντική πρόοδος σε όλη τη δέσμη μέτρων για τα αεροδρόμια. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε συμφωνία μια και οι θέσει Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου είναι πάρα πολύ κοντά. Στις χερσαίες μεταφορές μέσα στην εξάμηνη προεδρία μας πετύχαμε σημαντική πρόοδο τόσο στους ταχογράφους όσο και στους τεχνικούς ελέγχους οχημάτων. Οπωσδήποτε εκτιμώ ότι η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχίσει και θα συνεχίσει επί της Ιρλανδικής Προεδρίας. Στη γενική προσέγγιση για τον τραχογράφο σεβαστήκαμε την πλειοψηφία των κρατών μελών, ειδικά για το θέμα των οχημάτων 2,8 τόνων μέχρι 3,5 τόνων υπήρχε ομοφωνία στο Συμβούλιο για εξαίρεση. Δεν έχει να κάνει με το δικό μας εθνικό ενδιαφέρον ή όχι, δεν παρουσιάστηκε οποιαδήποτε πρωτοβουλία από την Επιτροπή στη διάρκεια του εξαμήνου μας. Έχω πληροφορηθεί ότι η νέα νομοθετική δέσμη τώρα θα παρουσιαστεί και θα εξεταστεί στο Συμβούλιο και η αναφορά γίνεται για το σιδηροδρομικό πακέτο το τέταρτο. Οι υποδομές στον τομέα των μεταφορών είναι εξαιρετική σημασία. Οπωσδήποτε οι επόμενοι μήνες θα είναι σημαντικοί και το Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να εργαστούν με επικοδομητικό πνεύμα για να επιτύχουν συμφωνία. Το θέμα των εκπομπών αερίων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ελπίζουμε ότι σύντομα θα εξευρεθεί λύση σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα, μέσω του Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας ΑΚΕΟ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για τον χρόνο τον οποίο έχετε αφιερώσει σε εμάς. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την ε, εργασία που επιτελέσατε ως προεδρεύων σε όλα τα θέματα που αφορούν τις μεταφορές. Χειριστήκατε φακέλους πολλούς σημαντικούς. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό και Ξέρω ότι θα συνεχίσετε να παρακολουθείτε και την εξέλιξη των φακέλων αυτών και κατά τη διάρκεια τη Ιρλανδικής Προεδρία. Εξ λοιπόν όλων των μελών της Επιτροπής μας και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Τι συνάδελφοι του ΕΛΚΑ. Εξ ονόματός σας έχω την ευχαρίστηση που δεχθώ τον ε, Ιρλανδό Υπουργό Μεταφορών της Ιρλανδίας και Προεδρεύοντα, τον κύριο Λέο Βαρατκάρ, ο οποίος θα μας εκθέσει τις θέσεις και τα θέματα ενδιαφέροντος της Ιρλανδικής Προεδρίας. Θα τον ακούσουμε πρώτα απ' όλα και μετά θα δώσω το λόγο στους συντονιστές για το λόγο και θα πρέπει να είμαστε όλοι σύντομοι να σεβαστούμε το χρόνο που μας έχει δοθεί. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για τη δυνατότητα που μου δίνει να παρουσιάσουμε τις προτεραιότητες της Ατλαντικής Προεδρίας όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον Κύπριο συνάδελφο Ευθύμιο για την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει ο ίδιος και η ομάδα του όσον αφορά τα πολύ σημαντικά ζητήματα στον τομέα των μεταφορών, ιδίως όσον αφορά την πολιτική των θαλασσίων μεταφορών, η οποία γνωρίζω ότι είναι προσφυλή σε πολλά άτομα της Επιτροπής αυτής. Είχα τη δυνατότητα να συναντηθώ με τον Μπράιαν, καθώ επίση και με πολλά μέλη τη Επιτροπή αυτή στο παρελθόν, καθώ προετοιμαζόμασταν για την Προεδρία μα. Και νομίζω ότι οι επαφέ αυτέ μου δώσαν τη δυνατότητα να καταλάβω καλύτερα ποιε είναι οι προτεραιότητε και ανησυχίε των μελών τη Επιτροπή αυτή όσον αφορά το ζήτημα των μεταφορών και του τουρισμού στην Ευρώπη. Όπω οποιοδήποτε δημοκρατικό οργανισμό, έτσι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί ένα μεγάλο φάσμα απόψεων και δεν αποτελεί βέβαια εξαίρεση η Επιτροπή αυτή. Αυτό όμω το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε προετοιμαζόμενο για την Ευρωπαϊκή Προεδρία είναι το πόσο καλά γνωρίζετε τα ζητήματα των μεταφορών τόσο σε επίπεδο τεχνικό όσο και ω προ επιπτώσει που θα έχουν για τον Ευρωπαίο πολίτη. Θα προσπαθήσω λοιπόν να, να χρησιμοποιήσω τη γνώση σα αυτή προκειμένου η Προεδρία μα να είναι ιδιαίτερα επιτυχή στον τομέα των μεταφορών. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, αλλά είμαι σίγουρο ότι όλοι έχουμε κάποιου κοινού στόχου. Τρει είναι οι πιο σημαντικοί κατά την άποψή μου. Πρώτον, η Ευρώπη να καταφέρει να ανακτήσει την οικονομία τη και να εξηγιάνει τα δημοσιονομικά τη στοιχεία να δοθούν περισσότερε ευκαιρίε απασχόληση ιδίω για του νέου και τρίτον και πιο σημαντικό να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να εργαστούμε πιο επικοδομητικά προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών. Σταθερότητα, θέση εργασία και ανάπτυξη είναι τα βασικά ζητήματα τη Ιρλανδική Προεδρία. Και ακριβώ αυτέ είναι οι αρχέ που χρησιμοποίησαμε προκειμένου να κάνουμε μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων στην Ιρλανδική Προεδρία. Όσον αφορά όλε μα τι ε, πολιτικέ, στα πλαίσια τη Ιρλανδική Προεδρία θέλουμε να δημιουργηθούν οι απαραίτητε προποθέσει για να οδηγηθούμε σε σταθερότητα, θέσει απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ξέρω ότι συμμερίζεστε κι εσεί την άποψη αυτή και ξέρω ότι ξέρετε ότι οι μεταφορέ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα για την ανταγωνιστικότητα και επίση για την πλήρη εφαρμογή τη ενιαία αγορά. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι στα πλαίσια και των μεταφορών η βασική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και ενοποιημένου, ολοκληρωμένου δικτύου μεταφορών. Ξέρετε ότι ε, η δική μας τριάδα προεδριών είναι η τελευταία προτού λήξει η θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιέζει λοιπόν ιδιαίτερα ο χρόνος και δυστυχώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν λειτουργούν πάρα πολύ γρήγορα. Καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε πρόταση γίνει από τώρα και στο μέλλον δεν θα έχει πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να ολοκληρωθεί στα πλαίσια τη νομοθετική διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο εργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με του άλλου δύο εταίρου τη Προεδρία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα, προκειμένου να καταφέρουμε να πάρουμε αποφάσει το στομότερο δυνατό. Ο Αντιπρόεδρο Επίτροπο Κάλλα με εξασφάλισε ότι θα δούμε κάποιε πολύ σημαντικέ προτάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τέταρτη δέσμη μέτρων για τι δρομικέ μεταφορέ, μια νέα πρόταση για την καθαρή ενέργεια τη μεταφορέ, που είμαι σίγουρο θα θέσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη όσον αφορά τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και τέλο θα έχουμε και μια νέα πρόταση όσον αφορά το δικαιώματα των επιβατών σε αερομεταφορέ. Επίση, υπάρχουν πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα, πολλέ άλλε σημαντικέ προτάσει, οποίες οποίε θα δούμε κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου. Καταρχά, μια νέα πρόταση κανονισμού όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια τη Ναυσιπλοεία. Επίση, θα υπάρχει μια νέα πρόταση όσον αφορά την ασφάλεια του επιβατηγού πλοίου και επίσης θα έχουμε την επόμενη φάση της εφαρμογής του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Μια άλλη σημαντική προτεραιότητα είναι και αυτή προκειμένου να καταφέρουμε να κάνουμε πιο, πιο αποτελεσματικό τον τομέα των αερομεταφορών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλές προτεραιότητες και ελάχιστο χρόνο στη θέση μας. Βασική μου προτεραιότητα είναι να καταφέρουμε να συντονίσουμε σωστά την Προεδρία αυτή προκειμένου να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να επικεντρωθώ πραγματικά στα σημεία αυτά τα οποία ανέφερα και να λειτουργήσω ω διαμεσολαβητή προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο τα βασικά ζητήματα των τομέα μεταφορών. Δεν νομίζω όμω ότι θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία ως αυτός σκοπός. Νομίζω ότι πάρα πολύ συχνά κάποιες προτάσεις αποδυναμώνονται στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή και πολλές φορές θα ήταν πολύ καλύτερο να μην είχαμε τελικά την πρόταση αυτή. Ένα από τα βασικά σημεία τη δική μα Προεδρία είναι ότι δεν προσπαθούμε να προωθήσουμε τη δική μα την εθνική ατζέντα. Λειτουργούμε καθαρά ευρωπαϊκά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε να κάνουμε τι ευρωπαϊκέ υποδομέ μεταφορών κατάλληλε και πιο αποτελεσματικέ. Ω οικονομία ανοιχτού εμπορίου, η Ιρλανδία εξαρτάται πάρα πολύ από ένα αποτελεσματικό δίκτυο οδικό και σιδηροδρομικό στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώ επίση και σε άλλε περιοχέ τη Ευρώπη. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Καταλαβαίνετε ότι τα σημεία συμφόρηση, η έλλειψη διασυνδέσεων, η υπερβολική εσωτερικοί διοικητικοί έλεγχοι στους λιμένες λειτουργούν ανασταλτικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, η οποία όπως ξέρετε βασίζεται πάρα πολύ στις εξαγωγές. Οι εξαγωγές αυτές θα εξαρτηθούν πάρα πολύ από την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως τα σημεία συμφόρησης ή ενεπαρκείς διασυνδέσεις. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι δύο βασικά σημεία στην Ελλαδική Προεδρία θα είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών καθώς επίσης και διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Δεν μπορούμε εμεί ω Ιρλανδία να κάνουμε τι επενδύσει όπω κάναμε στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε επενδύσει, απλώ οι επενδύσει μα θα είναι πιο αποτελεσματικέ, πιο ευφυεί πλέον. Αυτό βρίσκεται πραγματικά στην καρδιά των Ευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και του CEF. Να καταφέρουμε να κάνουμε δηλαδή στοχευμένε αποτελεσματικέ επενδύσει εκεί που θα δημιουργήσουν πραγματικά ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επίση, θεωρούμε ότι ο ιδιωτικό τομέα μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου να κάνει τι απαραίτητε επενδύσει στι υποδομέ. Στα πλαίσια του προγράμματος Συνδέοντας την Ευρώπη θέλουμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όμως και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε μια επικοδομητική απόφαση. Δεν θα έλεγα ότι είναι εξασφαλισμένο προπολογισμό για το πρόγραμμα Συνδέοντα την Ευρώπη. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν πολύ σημαντικέ πιέσει ω προ τον προπολογισμό αυτό. Εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ω Προεδρεύων αλλά και σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό προπολογισμό για το CF και ξέρω ότι ο συναδελφό μου, Υπουργό Επικοινωνιών Πατ Rabbit, θα ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά την ενέργεια και τι τηλεπικοινωνίε το να καταφέρουμε να πετύχουμε μια γρήγορη απόφαση για ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνουν και κατάλληλε επενδύσει. Ξέρω ότι οι συγητέ για τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ο κύριο Κουμουτσάκο και ο κύριο Ισμαήλ Ερτούκ, θα συνεργαστούν πολύ καλά με το Συμβούλιο προκειμένου να επιτευχθεί μια πολύ καλή απόφαση. Το ίδιο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ισχύει και για τον κανονισμό γιατί ο κανονισμό αυτό πραγματικά θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά για τι επόμενε. Ε, επενδύσεις που θα γίνουν σε ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών. Ξέρω ότι θα χρειαστεί να γεφυρώσουμε διαφωνίες οι οποίες ενδεχομένως να υπάρχουν και να καταφέρουμε να πετύχουμε μία μακροπρόθεσμη συμφωνία η οποία θα καθορίσει τα επόμενα 40 χρόνια στα πλαίσια των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η δέσμη μέτρων για του αερολομένε επίση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξέρετε ότι το Συμβούλιο είχε εκφράσει την άποψή του για τι τρει πτυχέ του κανονισμού, θόρυβο, χρονοθυρίδε και υπηρεσίε εδάφου. Περιμένουμε τώρα να δούμε και ποια θα είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τι υπηρεσίε εδάφου. Ξέρω ότι υπάρχουν ιδιαίτερε δυσκολίε και ευαισθησίε ω προ αυτό. Ξέρω όμω ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εσά και δεν κάνω λάθο το συζητήσα και σήμερα το απόγευμα. Και ελπίζω το Κοινοβούλιο θα καταφέρει να βρει μια θετική λύση που θα μα επιτρέψει και εμά να ολοκληρώσουμε το ζήτημα αυτό. Αυτή τη στιγμή διευθετηθεί το ζήτημα των υπηρεσιών εδάφου. Θα συνεργαστώ με τον κύριο Τζομαρία Ουτζία, τον Άρθουρ Τζαζάντα, καθώ επίση και τον Γιώργο Λάικτφριντ, για να πετύχουμε το, το ιδανικό αποτέλεσμα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ξέρετε ότι η Ιρλανδία είναι νησιωτική χώρα με μια ισχυρή ναυτική παράδοση και θέλει να προωθήσει ιδιαίτερα τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι προωθείται η σύμβαση αυτή ακόμα περισσότερο μέσω των προτάσεων που έχω γίνει για το κράτος λιμένα και το κράτος σημαίας. Η Σύμβαση Ναυτική Εργασία θα αρχίσει να ισχύει από τον Αύγουστο του 2013 και πρέπει η Ευρώπη να είναι έτοιμη για τη σύμβαση αυτή. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από του Ευρωβουλευτέ να γνωρίσουν ότι η διαδικασία επικύρωση είναι μακροχρόνια για πολλά κράτη-μέλη. Η επικύρωση ουσιαστικά αντιστοιχεί στην αναθεώρηση μια ναυτιλιακή νομοθεσία 100 ετών περίπου. Ξέρω όμω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να πετύχουν τα χρονοδιογράμματα τα οποία έχουμε θέσει. Ο Μπράιαν και οι υπόλοιποι στην Επιτροπή αυτή ξέρω ότι θέλουν να προωθήσουν πάρα πολύ τον, την εργασία που θα γίνει για το κράτος λιμένα, καθώ επίση και το κράτο σημαία, με το οποίο θα ασχοληθεί κυρίω η Επιτροπή Απασχόληση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ο κανονισμό για το ταχογράφο. Συνάντησα την κυρία Σίλβια Αντριάννα Τικάου το Δεκέμβριο και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε μια καλή απόφαση και στι δύο πλευρέ, και στο Κοινοβούλιο δηλαδή και στο Συμβούλιο. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να συζητήσουμε επίση όρις ω ισότιμη εταίροι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε λεπτομερή συζήτηση σήμερα, ούτε πρόκειται να μιλήσουμε για κόκκινε γραμμέ ή διαπραγματεύσει. Πάντω, σα υπόσχομαι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να στεφτούν με επιτυχία όλα αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποιε μελλοντικέ προτάσει τώρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του τριμερούς διαλόγου όμω στι επαφέ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ προτάσει, τι οποίε θα ήθελα πραγματικά να αρχίσει να εξετάζει η Επιτροπή Μεταφορών. Καταρχά, η τέταρτη δέσμη μέτρων για, το... για τι ηλεκτρονικέ μεταφορέ. Το πακέτο αυτό θεωρείται μια πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα για την δεύτερη πράξη νέα αγορά και πραγματικά βρίσκεται στην πρώτη θέση στην ατζέντα του Συμβουλίου. Δεν θέλουμε να υπάρχουν περαιτέρω καθυστερήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη δημοσίευση αυτή τη ανακοίνωση. Το πακέτο αναφέρεται σε τεχνικά ζητήματα που αναφέρονται στο ζήτημα τη διαλειτουργικότητα και τη ασφάλεια, αλλά και σε κάποια ευαίσθητα ζητήματα όπω η πρόσβαση στην αγορά, καθώ επίση και η υποχρεώση παροχή δημοσίων. Πρέπει καταρχά να ασχοληθούμε με την τεχνική πτυχή του ζητήματο αυτού, του νομοθετικού αυτού φακέλου, προκειμένου προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα πλήρω ολοκληρωμένο συνδρομικό σύστημα στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα σε σχέση με τον φάκελο αυτό και θα πρέπει να τον μετωπίσουμε τη δέουσα προσοχή. Ξέρω επίση ότι σήμερα το βράδυ θα γίνει και μία εκδήλωση από την κοινότητα Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων στο ξενοδοχείο Renaissance και ελπίζω πραγματικά να έρθετε κι εσείς στην συνάντηση αυτή. Τώρα, όσον αφορά το τα δικαιώματα των επιβατών των ε, αεροπορικών εταιριών και αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να προστατεύσουμε του ε, επιβάτε, κυρίω όταν υπάρχουν ακυρώσει πτήσεων, καθυστερήσει πτήσεων ή άρνηση επιβίβαση. Στα πλαίσια επίση του Ευρωπαϊκού Έτου του Πολίτη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε το φάκελο αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για του Ευρωπαίου πολίτε. Επίσης, μια ακόμα πρόταση πολύ σημαντική είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθαρή ενέργεια της μεταφοράς. Πολύ σύντομα θα δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση αυτή. Ο Επίτροπος Κάλλας θέλει να προωθήσει την πρόταση αυτή, γιατί πραγματικά θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ανάπτυξη υποδομών φόρτωσης και τροφοδοσίας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα επικεντρωθούμε κατά αυτόν τον τρόπο περισσότερο στις υποδομές φόρτωσης και τροφοδοσίας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ένα τομέα πολύ σημαντικό για την Ιρλανδία και ελπίζω πραγματικά ότι θα υπάρχει μια πολύ θετική συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και των Υπουργών στο Συμβούλιο. Θεωρώ ότι πραγματικά μπορούμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή για την προώθηση των ζητημάτων αυτών, ιδίω στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών του Ιουνίου. Επίση, στα πλαίσια των θαλασσίων μεταφορών θα ασχοληθούμε με το ζήτημα τη ασφάλεια επιβατικού πλοίου Ξέρετε ότι έχει περάσει ένα χρόνο από το ατύχημα του Κώσταν Κοκόρδια την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα. Και το δεύτερο ζήτημα που θέλουμε να προωθήσουμε είναι η πρωτοβουλία για τη γαλάζια ζώνη, προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό άκθο για τι θαλάσσιε μεταφορέ μικρών αποστάσεων. Η Επιτροπή Μεταφορών επίση είναι καθήλυν αρμόδια επιτροπή για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ζήτημα με το οποίο ασχολείται το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Ιρλανδικό Υπουργείο ε, Εξωτερικών Σχέσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε πώς θα, πώς θα εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ακτογραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιστοιχεί σε 89.000 χιλιόμετρα. Επίσης, θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το ζήτημα των, του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς επίσης και της διαχείρισης των παρακτήων ζωνών. Τον Φεβρουάριο συγκεκριμένα θα έχουμε πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, θέλουμε να ξεκινήσουμε ως προς αυτό και διοργανικές διαβουλεύσεις. Υπάρχουν επίσης κάποια τεχνικά ζητήματα από τα οποία ελπίζουμε να με τα οποία ελπίζουμε να ασχοληθούμε στο Συμβούλιο. Θέλουμε επίσης μια καλύτερη ευθυγράμμιση για τον θαλάσσιο εξοπλισμό, τον εξοπλισμό των πλοίων δηλαδή, και θα έχουμε επίσης και μια οδηγία για τα σκάφη εναψυχής, καθώς επίσης και μια οδηγία για τον θόρυβο από τα χήματα που χρησιμοποιούν μηχανήματα, μηχανές, με Επίση, όσον αφορά του τεχνικού ελέγχου, ε, αν δεν κάνω λάθο αύριο έχετε σχεδιάσει μια ακρόαση για το ζήτημα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε και με τι δύο πτυχέ τη πρόταση αυτή, τόσο του περιοδικού ελέγχου, όσο επίση και του ελέγχου που γίνονται στο δρόμο, καθοδόν. Η Κυπριακή Προεδρία ασχολήθηκε εν μέρη με του περιοδικού ελέγχου και είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια τη δική μα προεδρία να έχουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα προκειμένου, να βελτιώσουμε τα επίπεδα ασφάλεια. Του επόμενου έξι μήνε ελπίζουμε να έχουμε μια τοποθέτηση του Συμβουλίου για τα άλλα δύο ζητήματα, προκειμένου η Λιθουανία να μπορέσει να ξεκινήσει με τη σειρά τη διαπραγματεύσει με τον κύριο Κούν, την κυρία Σενάλοβα και την κυρία Σαβισάρ Τούμαστα. Επίση, η οδική ασφάλεια αποτελεί πολύ σημαντική προτεραιότητα για την Ιρλανδία. Προφανώ ε, δεν έχουμε εμεί την ε, μόνη και μοναδική εμπειρογνωμοσύνη για το ζήτημα αυτό. Πάντω, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι μια σημαντική διάσκεψη για την οδική ασφάλεια θα γίνει στο Δουβλίνο κατά τη διάρκεια της δικής μας της προκειμένου να ασχοληθούμε το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Θα ασχοληθούμε πιο ιδιαίτερα με τους σοβαρούς τραυματισμούς και η διάσκεψη αυτή θα γίνει στις 28 Μαρτίου στο κάστρο του Δουβλίνου θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε και εμεί ω ε, Ιρλανδική Προεδρία σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα τη πρόληψη των τραυματισμών και των ατυχημάτων. Επίση, η Ιρλανδία θα διοργανώσει την ένατη Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τεφή συστήματα μεταφορών από 4 έως 7 Ιουνίου του 2013, όπου θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε περισσότερο στα ωφέλη των ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Άλαν Κέλλη, ο οποίος είναι και πρώην δικό σας συνάδελφος, ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ζήτημα αυτό. Θέλω να αναφερθώ σε ένα ακόμα ζήτημα πολύ σημαντικό και για σας και για μένα, τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομίας, μπορεί πραγματικά να προωθήσει την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη παντού στην Ευρώπη. Ιδίως για τις περιοχές εκείνες και τις κοινότητες εκείνες που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλε οικονομικές ευκαιρίες και δυνατότητες. Η Ιρλανδική Προεδρία υποστηρίζει ιδιαίτερα τον σημαντικό αυτό ρόλο που μπορεί να δραματίσει ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν να ασχοληθούμε με όλες σχετικές με τον τουρισμό προτάσεις. Ιδίως θα αναφερθούμε στο πρόγραμμα COSME, ο οποίος αναγνωρίζει ιδιαίτερα την σημασία του τομέα του τουρισμού για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για τη δημιουργία μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης. Ο συναδελφός μου, ο κύριος Ρίτσαρτ Μπρέτον, ο οποίος είναι υπουργό Απασχόλησης, θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ζήτημα αυτό. Να αναφερθώ επίσης στην Task Force για τον τουρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικεφαλής είναι ο κύριος Κάρλο Φιντάντσα. Παρακολουθώ εκ του σύνεγγυ ε, τι δραστηριότητε τη της ε, Task Force αυτής. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι ο συναδελφός μου Jim Higgins, που προέρχεται από την ίδια χώρα με μένα, θα συμβάλλει πολύ σε αυτή την Task Force με τη δική του την εμπειρογνωμοσύνη. Ε, είναι ιδιαίτερα παθιασμένος με το ζήτημα του τουρισμού, ιδίως όσον αφορά την ε, Δυτική Ιρλανδία. Ο τουρισμός, ο πολιτιστικός, καθώς επίσης και αυτός που συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός. Ο, Ευρωπα... ο Ιρλανδικός Οργανισμός Τουρισμού θα διοργανώσει 27... 25 με Απριλίου μια σημαντική διάσκεψη στο κάστρο του Δουβλίνου όσον αφορά τον τουρισμό. Θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το ζήτημα του πολιτιστικού ε, τουρισμού και θα ήθελα επίση να καλέσω τα μέλη της Επιτροπής αυτής και ιδιαίτερα της Task Force να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνδιάσκεψη. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθώ σε μια άλλη πολύ σημαντική πρωτοβουλία που θα λαμβάνει χώρα στην Ιρλανδία το 2013 και αναφέρομαι στην πρωτοβουλία, στην εκδήλωση μάλλον The Gathering Ireland. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διάσκεψη που έχει ως στόχο να προωθήσει την Ιρλανδία, τους Ιρλανδούς, την πολιτιστική κληρονομιά της Ιρλανδίας, την ε, γαστρονομική της κληρονομιά, την γλώσσα, τον πολιτισμό. Σας προσκαλούμε λοιπόν να λάβετε κι εσείς ε, μέρος στην εκδήλωση αυτή που θα διοργανωθεί κατά τη διάρκεια του 2013. Σας προτείνουμε λοιπόν όσοι συμμετάσχετε μια πρώτη φορά επαγγελματικά σε κάποιες ε, συνδιασκέψεις μας να επανέλθετε κατά το δεύτερο ήμιση της Προεδρίας μας για να συμμετάσχετε και σε αυτή την εκδήλωση. Σας ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα, σίγουρα έχουμε πάρα πολλές προτεραιότητες και πάρα πολλή δουλειά την οποία πρέπει να επιτελέσουμε. Η επιτυχία μας θα, θα εξαρτηθεί από την πολύ επικοδομητική συνεργασία, την οποία είμαι σίγουρο ότι θα εξασφαλίσουμε. Είναι περιορισμένος ο χρόνος, προσβλέπω πραγματικά στις δικές ερωτήσει ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Δεδομένου ότι πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο, θα αρχίσω με τους συντονιστές. Τους παρακαλώ εκ των προτέρων να μην ξεπεράσουν τα τέσσερα λεπτά για να μπορέσουμε να σεβαστούμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Σύντομα και καθαρά ό,τι έχετε να πείτε λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Πρόεδρο της ε, του Συμβουλίου. Το πρόγραμμά σας είναι θαραλέο και πολύ ενθουσιώδες και ε, πραγματικά και εγώ είμαι από, μικρός, ε, από μικρή χώρα και οι εκπρόσωποι των μικρών χωρών συνήθως έχουν ε, το έθιμο να προωθούν επιτυχημένα τα ντοσιέ τους, τα θέματα τους. Το ΕΛΚ θα είναι στο πλάι σας σε πολύ σημαντικά θέματα έτσι ώστε να μην έχουμε απλώς μία ένα άθροισμα των εθνικών ε, ε, ευχών στη δουλειά που κάνετε. Από την πλευρά μας, ε, πολύ σημαντικό είναι το θέμα της γέφυρας μεταξύ της τεχνολογίας και των μεταφορών, οι πολίτες και οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίζουν την ε, προστιθέμενη αξία, να μην είναι μια Ευρώπη των βασάνων, αλλά της προστιθέμενης αξίας της ασφάλειας. Και αυτό ισχύει για αυτό το θέμα, για αυτό το φάκελο που ε, πραγματικά αφορά όλους τους πολίτες στις διάφορες μορφές μεταφορών. Έχουμε διάφορα ντοσιά που έχουμε ετοιμάσει για αυτό το θέμα και πολλέ πρωτοβουλίε που μπορούμε να επιδείξουμε για την προστιθέμενη αξία ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πολλά ζεστά καυτά θέματα. Στο πακέτο της αεροπορίας, ας πούμε, θα πάει πίσω στην Κομισιόν το θέμα, αλλά πρέπει και εδώ συνολικά να έχουμε με τη βοήθειά σας την προστιθέμενη αξία που χρειάζεται και το νέο πακέτο που θα έρθει. Ε, έχουμε ένα καλό παράδειγμα του τι, του τι περιμένουμε ως κοινοβούλιο. Θέλουμε τεχνολογικά πρώτον ε, γρήγορη πρόοδο, έτσι ώστε να έχουμε ένα σωστό και σημαντικό χώρο συνδρομικό για την Ευρώπη και από την άλλη να μην χαθούμε σε δογματικές ε, συζητήσεις για το άνοιγμα των, αγορών, των αγορών, τη δομή των ε, κοινωνιών της υπηρεσίας κτλ. Γιατί πρέπει ε, η αποτελεσματικότητα να είναι πιο σημαντική από το δέγμα το θεωρητικό που χρησιμοποιούμε στις συζητήσεις μας. Μόνο τότε θα έχουμε προστιθέμενη αρξία. Θα αφήσω και τους άλλους συναδέλφους να μιλήσουν για αυτό το θέμα, αλλά να μιλήσω πρώτα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τη χρηματοδότηση. Αν δούμε πώς πάει ε, το θέμα στο Συμβούλιο με τα χρηματοδοτικά μέσα, ε, βλέπουμε αυτή την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με δύο τρόπους. Ε, από τη μία έχουμε την επιτυχία και από την άλλη πραγματική αλληλεγγύη. Είναι σημαντικό τα διευρωπαϊκά δίκτυα πραγματικά να αποτελέσουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να ε, δοθεί έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας έτσι ώστε να έχουμε ένα εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση και συγκεκριμένες ε, περιφέρειες να έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Αν όμως συζητάμε και εδώ όπως και στις άλλες, ε, στους άλλους τομείς, μείον 5, μείον 6, μείον 30% δεν γίνεται τίποτα. Πείτε στους συναδέλφους ότι πρέπει να σβήνουμε μόνο project και όχι 10% από ένα project. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε ε, να χρησιμοποιηθεί σωστά το θέμα των διευρωπαϊκών ε, δικτύων και το χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για τη δική σας Προεδρία, αλλά συνολικά για τον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτά περιμένουμε από εσά τους επόμενους μήνες. Να ξέρετε ότι εμείς ως Κοινοβούλιο είμαστε στο πλευρό σας, όπως ήμασταν ε, και στο παρελθόν στα διάφορα θέματα, σύμφωνα με την Κομισιόν. Να πείτε όμως και στους συναδέλφους ότι αν ε, μπορεί το 1% από κάθε προϋπολογισμό, κάθε κρατικό προϋπολογισμό να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πραγματικά ε, θα μας βοηθήσει. Το θέμα είναι τι κάνουν οι χώρες με το υπόλοιπο 99% του προϋπολογισμού. Αυτό ε, είναι ένα θέμα, αλλά επίσης και το θέμα των Connecting Europe Facility πρέπει να μείνει ως έχει. Δεν πρέπει να υπάρχουν μειώσεις σε αυτό. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ελκαντράουι. εκ μέρους των Σοσιαλιστικής Ομάδας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την έκθεσή του. Καλή επιτυχία σας εύχομαι για την Προεδρία. Μας είπατε ότι η φιλοδοξία σας είναι να κάνετε καλή νομοθεσία ώστε οι εξαιρεσει και τα, όλα αυτά τα opt-out να μην λάβουν χώρα. Ναι, καλό είναι να κάνετε κοινοτική νομοθεσία, αλλά θα πρέπει και να εφαρμοστεί. Αυτό θα πρέπει να προσθέσετε, να θεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία. Τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να μπλοκάρουν κάποια θέματα. Στις αρχές Δεκεμβρίου έπρεπε να υπάρξει μια κάποια πρόοδος. Δεν επιτεύχθηκε όμως. Εκφράζουμε τη λύπη μας. Υπάρχουν πολλοί φάκελοι ακόμη παρεμφερείς που δεν έχουν προχωρήσει. Και πολλά παραδείγματα θα μπορούσα να αναφέρω όπου έχουμε συμφωνία, το σχετικό έγγραφο, τη σχετική νομοθεσία, αλλά τίποτε στην πράξη. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσετε να συνεισφέρετε σε αυτό. Αναφέρατε μία σειρά προτάσεων όπως το πακέτο των ε, σιδηροδρομικών μεταφορών που είναι πολύ σημαντικό και αναμένουμε και παρακολουθούμε εκ του σύναγγης και με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις. Η ομάδα μου πιστεύει ότι η αγορά είναι σημαντική αλλά δεν είναι και η πανάκια. Θα πρέπει η τεχνική διαλειτουργικότητα να εξασφαλιστεί επίσης και θα πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν και την κατάλληλη κατάρτιση να εργάζονται με καλές συνθήκες και κυρίως στον σιδηροδρομικό ε, τομέα των μεταφορών θα πρέπει οι εργαζόμενοι να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την, την δημόσια υπηρεσία επίσης να την ε, διασφαλίσουμε. Θα παρακολουθούμε λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγάλη προσοχή την εξέλιξη όλων αυτών των φακέλων. Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο θέματα. Στους ε, ψηφιακούς ταχογράφους που είναι ένα θέμα το οποίο ακόμη συζητείται και κάποιοι συνάδελφοι θα λάβουν το λόγο εκ των υστέρων ώστε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια στις οδικές μεταφορές, αλλά θα πρέπει να γίνονται και σεβαστοί από όλους οι κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, ώστε να έχουμε μια συνεκτική και εναρμονισμένη πολιτική οδικών μεταφορών. Οι κανόνες λοιπόν θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί και θα πρέπει να είμαστε και κατά του dumping, του κοινωνικού και των δυσκολιών που μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιοι, που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιοι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό. Τώρα όσον αφορά το ΣΕΦ, τη διευκόλυνση και τα δέδε στον τομέα των μεταφορών είναι δύο σημαντικά θέματα, αλληλένδετα μεταξύ τους, αλληλοεπηρεάζει το ένα το άλλο, αλλά το να αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια αν δεν έχουμε στο τέλος τα κατάλληλα μέσα για να τα θέσουμε σε εφαρμογή, δεν μας ωφελεί και πολύ. Οι φήμες δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξε στον τομέα αυτό. Δεν είναι πολύ ρόδινη η κατάσταση. Δυστυχώς, από ό,τι ακούσαμε, θα μειωθούν τα προβλεπόμενα κονδύλια. Σας ζητούμε λοιπόν εξ ονόματος της ομάδας μας να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το θέμα αυτό, ώστε να εξασφαλιστούν τα κατάλληλα κονδύλια, να μην μειωθεί η κοινοτική χρηματοδότηση. Υπολογίζουμε λοιπόν στην δική σας υποστήριξη ως Υπουργού Μεταφορών, ώστε να ασκήσετε πιέσει στους συναδέλφους σας, καθώς και στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στα επίπεδα Συμβουλίου και να τονίσετε κυρίως ε, την διάσταση ανάπτυξης, που άπτεστε της σωστής ε, ανάπτυξης του τομέα αυτού. Σας ευχαριστούμε κύριο Κατράου. Η κυρία Μάισνερ, εξ ονόματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε ε, Κύριε Υπουργέ, καταρχάς όταν μας παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας χάρηκα γιατί είδα ότι θα είναι μια καλή προεδρία όπως είναι ωραία και η Ιρλανδία ως χώρα. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα ε, σχετικά με το υγρό στοιχεία. Ε, η, Ιρλανδία όπως και η Κύπρος είναι ένα νησιωτικό κράτος και υπάρχουν πολλά θέματα που με τα οποία ασχολούμαστε τώρα όπως είναι η ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα. Υπάρχει αυτή η διακήρυξη της Λεμεσού ε, κατάλαβα από την προηγούμενη ομιλία ότι θα τη συνεχίσετε. Υπάρχει και ο κανονισμός ε, για τον ε, θαλάσσιο χώρο. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με αυτά και ελπίζω ότι θα έχετε μια καλή συνεργασία και είμαι πεπισμένη ότι αυτό το σχέδιο της μπλε ανάπτυξης θα είναι ένα καλό πρόγραμμα. Επίσης όσον αφορά τον ILO Θεωρώ ότι έχουμε συμφωνήσει πως αυτό είναι σημαντικό. Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να κυρωθούν. Είπατε ότι θέλετε να δράσετε ως διαμεσολαβητής και να προωθήσετε στο μεταξύ και μία εθνική ατζέντα. Ε, είναι καλό αυτό, ελπίζω πραγματικά να επηρεάσετε θετικά και τα άλλα κράτη-μέλη ώστε να υπάρχει κύρωση. Ένα τελευταίο θέμα σχετικά με τα θαλάσσια. Μιλήσατε για την ασφάλεια των επιβατών. Ε, υπάρχει το ατύχημα του Κώστα Κονκόρντια και πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα που υπάρχει στην Κομισιόν. Ε, το Φλαμίνια δεν το αναφέρατε ήταν ένα γερμανικό ε, πλοίο, όμως αυτό μπορούμε να δούμε ε, ήδη από φέτος το καλοκαίρι ότι ε, αυτό το σύστημα που έχουμε για έκτακτη ανάγκη στα λιμάνια δεν λειτουργεί. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια πρόοδος και σε αυτό το θέμα. Τώρα, για άλλους τομείς, το σιδηροδρομικό πακέτο για παράδειγμα, είμαι από την Γερμανία η οποία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο Επίτροπος λέει ότι είναι η Γερμανία ενάντια του υπόλοιπου κόσμου. Για μένα είναι σημαντικό να δούμε τι είναι πρακτικό σε επίπεδο και ανταγωνισμού, αλλά αυτό έχει να κάνει ε, όχι μόνο με το από ποια χώρα προερχόμαστε. Μιλήσατε για τον τους ευρωπαϊκούς ουρανούς, τον ενιαίο εναέριο χώρο. Χαίρομαι που θέλετε να επιτύχετε πρόοδος διαμεσολαβητής, ειδικότερα στο ΦΑΜΠΕΚ στον ενδιάμεσο ένα αέριο χώρο της Γαλλίας και της Γερμανίας όπου δεν έχει γίνει καμία πρόοδος. Αν το καταφέρετε αυτό ως διαμεσολευητής πραγματικά θα είναι εξαίρετο και σας ε, εύχομαι κάθε τύχη. Μακάρι να γίνει. Δεύτερη, τώρα μια άλλη ε, ένας άλλος τομέας, η ψηφιακή ταχογράφη, συμφωνώ με τον συνάδελφο Γκρός, έχει να κάνει με την ασφάλεια ε, των μεταφορών, αλλά έχει να κάνει και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες όλο και περισσότερο ε, αναφέρονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όμως ε, βλάπτονται και από τη γραφειοκρατία η ασφάλεια είναι το ένα κομμάτι, αλλά και η γραφειοκρατία είναι το άλλο. Πρέπει να τα προσέχουμε στη οδηγίες μας. Και το τελευταίο, που είναι ένα σημαντικό project, τα TNT, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το SEF, Connecting Europe Facility. Από το 2009 που είμαι στο Κοινοβούλιο, ποτέ δεν είχα βιώσει να υποστηρίζουν όλα τα κόμματα ε, ένα τέτοιο θέμα όπου η Ευρώπη αναφέρεται ως ένας ενιαίος χώρος και υπάρχει και αντίστοιχη χρηματοδότηση. Από την πλευρά του Κοινοβουλίου πραγματικά θα προσπαθήσουμε σε επίπεδο χρηματοδότησης τουλάχιστον να κρατήσουμε τα πράγματα ως έχουν. Το Συμβούλιο φέρει, θέλει φυσικά να μειώσει κάποια πράγματα, αλλά χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια κοινή ε, ε, θέση και εσείς ως Προεδρία πρέπει να έχετε τα μάτια σας στα πιλωτικά ε, προγράμματα τα οποία θα μπορούν να γεννήσουν χρήματα και να μπορέσουμε έτσι να χρηματοδοτήσουμε ακόμα και τον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Προεδρεύοντα και σας εύχομαι καλή τύχη. Σας ευχαριστούμε κυρία Μάισνερ. Ο κύριος Τσίλερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό και γενικότερα την Ιρλανδική Προεδρία για το πολύ καλά δομημένο πρόγραμμα το οποίο έχουν παρουσιάσει. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα την τέταρτη δέσμη μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Εσείς εκπροσωπώντας την Ιρλανδία σε συνεργασία με την Λιθουανία και την Ελλάδα, τις επόμενες δηλαδή προεδρίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθείτε με το ζήτημα των σιδηροδρόμων. Θα πρέπει όλος ιδιαίτερος να ασχοληθείτε με την ιδιαίτερη κατάσταση εκείνων των χωρών που δεν τυχαίνουν πολύ καλής κατανόησης ε, από τις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Μία συγκεκριμένη ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Είπατε ότι θέλετε να ξεκινήσετε με την τεχνική πτυχή, δηλαδή με, το, με τα πιστοποιητικά, τα τεχνικά, και στη συνέχεια θα αφήσετε από ό,τι φαίνεται τα πολιτικά ζητήματα για μια αργότερη εξέταση κάποια στιγμή στο μέλλον. Ανησυχώ όμω πρόκειται πραγματικά να διαχωρίσετε την δέσμη μέτρων, δηλαδή ζήματα αποσύνδεσης και απελευθέρωσης θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της επόμενης νομοθετικής θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τώρα την διευκόλυνση συνδέοντας, την Ευρώπη και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, προφανώς και τα δύο ζητήματα αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Ελπίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή επιτευχθεί μια απόφαση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα μπορέσουμε από κοινού να καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τις κατευθυντήρες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Και ελπίζω ότι θα είστε πάρα πολύ αυστηροί όσον αφορά την επιλογή των σχεδίων, των προγραμμάτων που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν, δεδομένου μάλιστα και του περιορισμού που υπάρχει στα κονδύλια. Και μία ακόμα ερώτηση από μένα που προέρχομαι από μία χώρα συνοχής. Θα ήθελα να συζητήσω να προσπαθήσετε να εξασφαλίσετε και να διατηρήσετε τη χρηματοδότηση για τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη και να διατηρήσετε γενικότερα τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής στα επίπεδα του παρελθόντος. Αν η χρηματοδότηση αυτή μειωθεί, τότε οι χώρες της πολιτικής συνοχής δεν θα καταφέρουν να κάνουν σπουδαία πράγματα. Όσον αφορά τώρα το πακέτο ασφάλειας για τις θαλάσσιες μεταφορές. αν λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση με το Κώστα Κονκόρντια και την διερεύνηση του ατυχήματος που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και το πώς ασχολούνται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το ζήτημα αυτό, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την νομοθετική πρόταση για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων. Θα καταφέρουμε να αποδείξουμε κατά αυτόν τον τρόπο ότι μπορούμε στην Ευρώπη να βελτιώνουμε τις συνθήκες ασφάλειας γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε εξ ονόματος των Πρασίνων, κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και σας εύχομαι καλή τύχη φυσικά. Έχω σημειώσει κάποια θέματα, τα δικαιώματα των επιβατών πάντοτε ακούγεται καλό. Ε, υπάρχει μια ανεξάρτητη ε, ε, αρχή διαμεσολάβησης για τα ε, αεροδρόμια, γιατί είναι πολύ δύσκολο κανείς να βρει, να βρει κάπου να ε, διαμαρτυρηθεί. Πάντοτε στα δικαστήρια μπλοκάρονται τα θέματα. Τελευταία στιγμή, ε, όταν υπάρχει θέμα διατησίας, ε, δεν προχωρεί. Το ίδιο λοιπόν που υπάρχει στην αεροπορία καλό θα ήταν να έχουμε και στους σιδηροδρόμους. Δεύτερον, πρέπει να επενδύσουμε πιο έξυπνα είπατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που το είπατε αυτό. Δεν υπόθηκε αλλού, όμως εγώ το λέω, ως τώρα έχουμε επενδύσει χαζά και με λιγο, λιγότερη ευφύεια. Έχουμε πράγματα που δεν έχουμε επιτύχει στον ευρωπαϊκό χώρο. Και ε, έχουμε δει ότι υπάρχουν δυσκολίες. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα στην Ευρώπη για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά μια άλλη πολιτική. Ε, χρειαζόμαστε άλλα σημεία βασικά. Και ό,τι και να γίνει, όσα και χρήματα και αν κόψει το Συμβούλιο, δεν... Ε, όποια ε, και αν είναι τα project που θα σβηστούν, ε, πάντοτε ε, λείπουν χρήματα. Ας πούμε, στην ε, ε, Γερμανία έχουμε ε, την σύνδεση ε, Βερολίνο-Μπρεσλάου που κοστίζει 300 εκατομμύρια και δεν, μπορεί να, δεν μπορούν να δοθούν ενώ υπάρχουν μεγαλύτερα project που ε, μπορεί να κοστίζουν περισσότερο και να μην δίνονται. Και να δίνονται, συγγνώμη. Τα πράγματα δηλαδή μετά τον πόλεμο είναι χειρότερα από ό,τι πριν. Άρα καλό θα ήταν να επενδύουμε πιο ε, έξυπνα έτσι ώστε οι επόμενες και μεθεπόμενες ε, γενιές να έχουν τις ε, θετικές επιπτώσεις. Μέχρι το τέλος του 2012 θα υπάρχει χαλάρωση, είπατε, για το θέμα των ταχογράφων. Επίσης, πάντοτε αμφιβάλλω για το λόγο της Κομισιόν. Ήταν στην αρχή ο Γενάρης, μετά τώρα είναι Φλεβάρης, μετά ίσως να έρθει ο Μάρτης. Ποια είναι η δική σας θέση. Καθαρή ενέργεια, το είπατε. Έχουμε τον στόχο μείωσης κατά 20% των εκπομπών μέχρι το 2020 και να γίνουμε κατά 20% πιο αποδετικοί. Στο μεταξύ, οι αεροπορικές μεταφορές και οι εκπομπές στη στρατόσφαιρα είναι πέντε φορές μεγαλύτερες από ό,τι στο έδαφος. Μιλήσαμε για, τους, για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Στο Ζαρμπρούκεν ε, υπάρχουν επιδοτήσεις 5,5 εκατομμύρια ευρώ για το αεροδρόμιο. Στο Κάσελ υπάρχει ένα αεροδρόμιο για ε, αεροπορικές εταιρείες που είναι αφαιρέγγες και έχουν ε, δράση μόνο στον τομέα της αναψυχής. Εσείς είστε έτοιμοι να σβήσετε αυτές τις ε, υπερβάλλουσες δαπάνες ε, και να ε, βγάλετε από το χάρτη αυτά τα αεροδρόμια που δεν έχουν καμία λειτουργία. Για το κόστο Concordia και άλλα αντίστοιχα θέματα που αναφέρθηκαν υπάρχει κάποια συζήτηση στο Συμβούλιο. Γιατί όταν έρχεται το θέμα πάντοτε όλα τα κράτη που σχετίζονται με το θέμα πάντοτε κοιτάνε την εθνική τους πλευρά και πραγματικά εδώ όλοι θεωρούμε ότι αυτό δεν πρέπει να ισχύει. Όταν υπάρχει ανάγκη, η εθνική διάσταση δεν πρέπει να παίζει ρόλο. Για τις υπηρεσίες εδάφους, ξέρετε την πλειοψηφία με την οποία απορρίφθηκε το θέμα στο Κοινοβούλιο. Το ερώτημά μου, θεωρείται λογικό εμείς να έχουμε κάποιον ευρωπαϊκό κανονισμό που θα είναι σχετικός ε, μόνο για τρία ή τέσσερα αεροδρόμια στα επόμενα 10-15 χρόνια. Γιατί για τέτοιες λεπτομέρειες κάνουμε ευρωπαϊκούς νόμους όταν ξέρουμε ότι αυτοί που φτιάχνουν τους νόμους ποτέ δεν τους στηρούν τελικά. Όπως έγινε με τους ανοιχτούς ουρανούς. Την 5η Δεκεμβρίου έπρεπε να είναι έτοιμα τα FAPS για να μπορέσουμε να κερδίσουμε σε εκπομπές, σε χρήματα και σε χρόνο. Σε μια κατάσταση win-win που θα κερδίζουν όλοι. Όμως το Συμβούλιο ο συνομοθέτης που τα υποστήριξε όλα, το αρνείται, λέει ότι εγώ κάνω τους νόμους μου, οι πολίτες πρέπει να τους ακολουθούν, αλλά εγώ όχι. Εγώ ε, στα γερμανικά θα το έλεγα, τους χέζω τους νόμους, αλλά αυτά δεν πρέπει να τα λέμε εδώ. Έχουμε ένα κράτος δικαίου στην Ευρώπη, αλλά ο καθένας αυθαίρετα από τα κράτη-μέλη τους ε, παραβιάζει. Για την ασφάλεια των μεταφορών ξέρουμε ότι ε, στους δρόμους γίνονται πολλά ατυχήματα λόγω μεγάλης, μεγάλης ταχύτητας. Πριν από 25-26 χρόνια έγινε ε, μια πρόταση της Κομισιόν για τη ρύθμιση της ταχύτητας ε, όπου ε, οι δήμοι και οι κοινότητες ε, θα έπρεπε να ρυθμίζουν από μόνες τους το τέμπο 30, δηλαδή πού θα οδηγεί κανείς και με ποια ταχύτητα. Στο Βερολίνο, για παράδειγμα, υπήρχε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν τώρα κάποιες πρωτοβουλίες των πολιτών και στην Ιρλανδία και στην Μεγάλη Βρετανία ε, υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Κάνετε κάτι. Όλοι έχουν όρια ταχύτητας. Στη Γερμανία όχι. Τι γίνεται ε, λοιπόν με αυτό το θέμα. Ε, θα υπάρχει ο καθένας να έχει τα δικά του όρια ή θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό ε, όριο σε 120 χιλιόμετρα για παράδειγμα. Εμείς είμαστε για τα 120 πέρα, αλλά εντάξει. 8 λεπτά μίλησε ο κύριος, πάρα πολύ. Μάλιστα. Θα πρέπει να τηρήσετε όμω παρακαλώ πολύ το χρόνο ομιλία, γιατί θα πρέπει να έχει και το χρόνο ο Υπουργό να απαντήσει στη συνέχεια. Ο κύριος Κόιτσεκ τώρα έχει το λόγο, εξ ονόματο της Γκούε. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι προτεραιότητε που μα παρουσίασε η Ιρλανδική Προεδρία είναι πολύ σημαντικέ Η οικονομική ανάπτυξη, θέσει απασχόληση, σταθερότητα, ανανέωση της εμπιστοσύνη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αν θέλουμε όμω πραγματικά να επιτύχουμε αυτού τους στόχους και αναφερθήκατε επίση και στον τουρισμό και αυτό το θεωρώ πολύ θετικό. Όντω πραγματικά ο τουρισμό δημιουργεί πάρα πολλέ θέσει εργασία παγκοσμίω. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, πρέπει να καταφέρουν να εντοπίσετε τα σημαντικότερα προβλήματα όσον αφορά τι οδικέ μεταφορέ. Μιλάμε ακόμα για τις υποδομέ, για την οδική ασφάλεια. Το βασικό όμω ζήτημα το οποίο πραγματικά μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την Ιρλανδική Προεδρία να εστιαστεί περισσότερο στην ε, ευθυγράμμιση των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την οδική ασφάλεια, όσον αφορά τώρα την δέσμη μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Το πρώτο πακέτο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Είναι μια απόλυτη καταστροφή και δεν αφορά μόνο αυτό την ε, γερμανική εταιρεία στυροδρόμων Θεωρώ ότι κυριαρχεί παντού στην Ευρώπη μια τεράστια σύγχυση και το μόνο που θα καταφέρουμε με την ελόγω νομοθεσία είναι να καταστρέψουμε τελικά τους σιδηροδρόμους στην ε, Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα τι εσωτερικέ πλωτέ μεταφορέ, καταλαβαίνω ότι ω Ιρλανδοί ενδιαφέρεστε περισσότερο για τι θαλάσσιε μεταφορέ. Η δική μου όμω χώρα περιβάλλεται τελικά από ξηρά και αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι εσωτερικέ πλωτέ μεταφορέ. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι ο πιο σημαντικό ποταμό για τι πλωτέ αυτέ μεταφορέ είναι ο δούναβη, όχι μόνο ο Ρήνο και η παραπόταμή του. Επομένω πρέπει να κάνετε κάτι σημαντικό και στην κεντρική Ευρώπη. Ας μην νομίζετε ότι ο Δούναβη βρίσκεται κάπου πέρα από τη βγαίνει και ότι ε, αφορά μόνο ελάχιστε χώρες. Αντίθετα, η σημασία του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν θέλουμε να αυξήσουμε την οδική ασφάλεια, νομίζω ότι ε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε κοινού κανόνε στην Ευρώπη και όσον αφορά τι αεροπορικέ μεταφορέ, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τι ενισχύσει. Υπάρχουν κάποιε εταιρείε, οι λεγόμενε low cost, όπω η Ryanair, που λειτουργούν και συμπεριφέρονται σαν καουμπόι σε ένα μπαρ, ουσιαστικά με ιδιαίτερη έπαρση θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε και σε αυτές τις εταιρείες να επιβάλλουμε κάποιους ελάχιστου κανόνες. Δεν έχω κάτι εναντίον τη εταιρεία αυτή, Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να μην ξεφεύγουν από του κανόνε. Αν δεν κάνω λάθο, υπάρχει μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει να κάνει με τα άτομα με ειδικέ ανάγκες στι αεροπορικές μεταφορές. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει κάποιε εταιρείε όπω και η Ryanair να συμμορφωθούν με του κανόνε που είχε εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, ασχολούμαι εμεί πάρα πολύ με, τις, με τα ατυχήματα, τα θαλάσσια ατυχήματα. Το Κώστα Κονκόρντια, το σχετικό ατύχημα, έλαβε χώρα πριν από ένα χρόνο. Είπατε ότι μία επιτροπή ερευνητική πρόκειται να συσταθεί σε ένα μήνα περίπου και σε ένα χρόνο θα έχουμε την τελική έκθεση. Ελπίζω η Ιρλανδική Προεδρία να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υποβληθεί τελικά η έκθεση αυτή για το Κώστα Κονκόρντια. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους αλλά όπως βλέπετε και εσείς έχουμε καθυστέρηση. Σας ε, ευχαριστώ λοιπόν εκ των προτέρων που δεν θα μακρηγορήσετε περισσότερο από δύο λεπτά ο καθένας. Δίδω το λόγο στον κύριο Βάνταλα. Voorzitter, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι που αναφέρατε το θέμα της ασφάλειας. Ιδιαιτέρως. Και θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για την ασφάλεια των εναερίων μεταφορών. Όπως ξέρετε, γίνονται πολλά για τους ε, πιλότους, πολλά διάβασα και ανησυχώ και πολύ. Κυρίως ε, οι ώρες ανάπαυσης, οι ώρες εργασίας των πιλότων, είναι ανησυχητικά όλα αυτά. Θα κάνετε κάτι, πιστεύετε για την ασφάλεια των αέριων μεταφορών ότι είναι αρκετός ο χρόνος ανάπαυση για τους πιλότους. Τώρα όσον αφορά τη Ryanair, πολύ λόγος γίνεται για αυτή την αεροπορική εταιρεία ίσως de jure και de facto σέβονται τους κανόνες. Αλλά υπάρχει μία κουλτούρα την οποία καλλιεργεί αυτή η εταιρεία, κυρίως όταν μπορεί να αποφασίσει ο υπεύθυνο πόσα καύσιμα θα φορτώσει στο αεροπλάνο ή όχι. Αυτό είναι από την οπτική γωνία της ασφάλειας. Σωστό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που είστε σύντομοι, η κυρία ευχαριστω σας ευχαριστω που ειστε συντομοι σε κυρια τσικαο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στην Ιρλανδική Προεδρία και να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την διαθεσιμότητά του και για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε όσον αφορά τον φάκελο που αφορά τους ψηφιακούς ταχογράφους. Δεν πρόκειται για ένα εύκολο φάκελο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν και εγώ μαζί με τους συναδέλφους, κυρίως με τον κύριο ε, διευθυντή τον κύριο Higgins, καλώς με τους συναδέλφους των άλλων πολιτικών ομάδων. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας τον φάκελο αυτό. Προφανώς Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε εκτενείς συναντήσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να διαπραγματευτούμε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ή πρέπει να ξέρετε ότι η βούλησή μας στην Επιτροπή Μεταφορών είναι να μπορέσουμε να, υλο... να ολοκληρωθεί η τη της Ελληνικής Προεδρίας το θέμα αυτό. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ και στην οδηγία που αφορά την ε, ενοποίηση των διπλωμάτων οδήγηση των επαγγελματιών οδηγών. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να καταλήξουν σε κοινή θέση και να ζητήσουν από την Επιτροπή να κάνει μελέτη επιπτώσεων και να αλλάξει την πρόταση που έχει υποβάλει ανάλογα με τα πορίσματα αυτής της μελέτης επιπτώσεων. Τώρα, για τους ε, ταχογράφους υπάρχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους αφορά η ενδεχόμενη συμφωνία στην οποία θα καταλήξουμε. Θα θέλαμε λοιπόν αυτό το θέμα να το μελετήσετε κατά προτεραιότητα. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρά όπως και οι άλλοι συνάδελφοι τον Υπουργό για την πολιτική βούληση και την φιλοδοξία του να προχωρεί στα πλαίσια αυτού του του πολύ φιλόδουξου προγράμματος, διότι η σταθερότητα, η ανάπτυξη και η θέση επασχόληση είναι σημαντικό θέμα. Όσον αφορά το τέταρτο πακέτο για τις συνδρομικές μεταφορές, θα ήθελα να ξέρω γιατί στις διάφορες προτάσεις δεν υπάρχει η κοινωνική διάσταση. Διαφορετικά, αυτά τα οποία θέλουμε να θεσπίσουμε δεν θα έχουν καμία ισορροπία. Είναι απαραίτητο λοιπόν για λόγους ισορροπίας να υπάρχει αυτή η κοινωνική ε, διάσταση. Τώρα, όσον αφορά τις εναέριες μεταφορές, δεν είναι τα θέματα τα οποία τις αφορούν πάρα πολύ ε, ικανοποιητικά και θα θέλαμε τα θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνική διάσταση να τα εκτάσει η Επιτροπή Επασχόληση. Τώρα, όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών των ε, αερίων ταφώνων, θα θέλαμε να γίνουν προτάσει εναρμόνιση. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα σήμερα δεν είναι ότι υπάρχουν κάποιε εταιρείε οι οποίε μεταχειρίζονται του επιβάτε, αλλά εμεί ω επιβάτε δεν ξέρουμε τι ακριβώ πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή: Θα κάνετε κάτι και για τους επιβάτες των πλοίων Τώρα, όσον αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, θα ήθελα να σας πω το εξής. Ε, στο όλο αυτό θέμα η Ισπανία και η Πορτογαλία μαζί είχαν προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά τώρα τελευταία υπήρξαν κάποιες διαφωνίες και θα ήθελα με την πολιτική σας βούληση να προχωρήσουν τα πράγματα. Στον τομέα του τουρισμού είπατε ότι δεν θα ασχοληθείς με το θέμα αυτό δεδομένου, λυπάμαι διότι για το θέμα αυτό έχετε πολύ σαφείς απόψεις, θα θέλαμε να υπάρχουν ε, τέτοιου είδους ε, ιδέες που θα τεθούν ε, σε εφαρμογή. Επίση είδα ότι εσείς ε, θα οργανώσετε σχετικά με το θέμα αυτό μια διάσκεψη του Δουβλίνο, θα συμμετάσχει στα θέματα οδικής ασφάλειας και των ε, σοβαρών τραυματισμών, αν το καθίσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας απασχολεί και θα μας απασχολεί και στο μέλλον. Και τελικά, στα πλαίσια των θεύτη ε, διευκόλυνση για την Ευρώπη, ε, σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία αυτή και θα συνεργαστούμε στα πλαίσια των δυνατήτων μα. Ευχαριστώ κύριος Κόχ. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, νομίζω ότι βρίσκεστε στο σωστό δρόμο, διότι αναγνωρίσατε ότι οι μεταφορές δεν είναι κάτι το οποίο ως πολιτική και ως τομέας λειτουργεί από μόνο του. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες και βεβαίως χωρίς μεταφορές δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ανάπτυξη, ούτε θέσεις επασχόλησης, ούτε ευημερία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για το φιλόδοξο πρόγραμμά σας. Όσον αφορά την βελτίωση της αποδοτικότητας, την σταθερότητα και την ανάπτυξη, έχετε την πλήρη η υποστήριξή μα. Η παρατήρηση μου, λέει ο πρόεδρο είναι ότι είναι πολύ πιο σύντομη οι κυρία συνάδελφοι από τι κυρίε συναδέλφου. Κύριο Χίγκη, ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, προεδρεύοντα για την παρουσία του και για τις προτεραιότητες που μας ανέφερε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Είπε ότι, ε, ο υπουργό ότι δεν, είμαστε, δεν έχουμε το μονοπόλιο στην Ιρλανδία για την οδική ασφάλεια. Αν δείτε του στόχου τους οποίου έχουμε θέση ε, από το 2001 τον στόχο μας δεν τον υλοποίησαμε στο 2010 να μειώσουμε τους ε, τραυματίες θάνατου. Ένας από τους το 1972 ε, 640 άτομα έχασαν ε, ε, τη ζωή τους μετά από πολλά χρόνια, 160. Ο στόχος μας όμως είναι να έχουμε μηδενικούς θανάτους, όπως η Σουηδία. Και νομίζω ότι στο Δουβλίνο η σχετική διάσκεψη που θα γίνει για την ασφάλεια το Μάρτιο είναι πάρα πολύ σημαντική. Κύριε Προεδρεύοντα, καλή τύχη για την Ιρλανδική Προεδρία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ερτού έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες. Σας ε, εύχομαι ότι καλύτερο για την Προεδρία. Να ζητήσω συγγνώμη που δεν ήμουν εξ αρχής ε, στην παρουσίασή σας ε, λόγω καθυστέρησης, όμως θα ήθελα να θίξω ένα σημαντικό θέμα που έχει να κάνει και πάλι με τα χρήματα. Φαίνεται ότι ε, στο πολιτές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο μας ε, ανέφεραν ότι υπάρχουν πολλά χρήματα, ειδικότερα όσον αφορά στο ΣΕΦ. Εξαρτιόμαστε λοιπόν από την χρηματοδότηση. Από τη μία, τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να προωθήσουν την πρόταση έτσι όπως την κατέθεσε η Κομισιόν και από την άλλη, αυτά τα σχέδια ε, για την ε, χρηματοδότηση ε, την χάνουν επιφυλάξεων. Έτσι λοιπόν έχουμε λιγότερα χρήματα και αυτό τελικά οδηγεί στο να μην έχουμε μια εξέλιξη όπως θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε κατά των διασυνοριακών ευρω... Ε, εμποδίων και πρέπει η διαλειτουργικότητα να λειτουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να έχουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω για άλλη μια φορά να μας ε, υποστηρίξετε σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Αρτού. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις και να κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση και να πω ότι το πρόγραμμά σας είναι πάρα πολύ συνεκτικό. Επίσης, να σας ευχαριστήσω ότι ήδη έχετε αρχίσει να συνεργάζεστε με κάποιους συναδέλφους για να ληφθούν αποφάσεις. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση. Έχετε ως προεδρεύον στον τομέα των μεταφορών να μας πείτε κάτι για την ε, χρηματοδότηση για τα ΔΕΒ ή θα ακολουθήσετε την Ιερική εδώ. Επίσης, είστε γιατρός εσείς. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε την Κομισιό να φέρει σε αίσιο πέρας ε, το τέταρτο πακέτο το σειροδρομικό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια που κάνατε και τις ερωτήσεις που κάνατε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσες περισσότερες μπορώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τα ευγενικά σας λόγια, για την υποστήριξή σας στην αρχή της Προεδρίας μας. Κύριε Γρός. μιλήσατε για τους ταχογράφους και συμφωνώ ότι το κλειδί εδώ είναι η προστιθέμενη αξία αυτό είναι ένα από του τομεί στον οποίο κατά διάρκεια τη Προεδρία μπορούμε να προχωρήσουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μπορούμε και να προσθέσουμε τις ε, εργαζόμενους και να εξασφαλίσουμε την οδική ασφάλεια. Πολύ όπως ο κύριος Τζον και ο Πρόεδρος, καθώς και άλλοι συνάδελφοί σας, ανέφεραν το ΣΕΦ και τα ΔΕΔ στον τομέα των μεταφορών. Ξέρουμε ότι πρόκειται για σημαντικά θέματα και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε τα κονδύλια που θέλουμε για να υπάρξει ανάπτυξη για την Ευρώπη, να κάνουμε επενδύσει, να εξασφαλίσουμε θέσεις απασχόλησης ώστε να κάνουμε έργα υποδομών και στον θέμα της, στον τομέα της ενέργειας. Και θα κάνω ό,τι μπορώ και στην Ιρλανδία αλλά όπως ξέρετε είμαι και ρεαλιστής. Όλες οι αποφάσεις δεν θα ληφθούν από μένα, αλλά σε ανώτερο επίπεδο. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε. Εάν μειωθούν τα κονδύλια και ο προπολογισμό, θα πρέπει να δούμε αυτά τα χρήματα που διαθέτουμε, πώς θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα προσπαθήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διαθεσή μας επίσης να τα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα κάνουμε εξιολογήσεις, όπως πρέπει. Η κυρία Μάισνερ και άλλοι συνάδελφοί της μίλησαν και για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ότι ήταν εξαιρετικά αργή η πρόοδος που επιτεύθηκε. Και είναι απογοητευτικό αυτό το θέμα. Διότι έχουμε ένα ενιαίο μάμισμα, μια ενιαία εσωτερική αγορά, αλλά δεν έχουμε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου των αερίων μεταφορών εξαιτία των πολυπλοκοτήτων που παρουσιάζονται. Η Επιτροπή είναι αυτή που θα αποφασίσει τι θα κάνει βεβαίω όσον αφορά την όλη διαδικασία, αλλά θα θέλαμε να προχωρήσει το όλο σχέδιο. Δεν ξέρω αν θα αρχίσει την ε, διαδικασία παραβάσεων η Επιτροπή. Όχι αυτό το θέμα. Το γεγονός ότι μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας ε, ε υπάρχει καλή συνεργασία όπως και μεταξύ Δανίας και Σουηδίας. Δεν ξέρω αν τα θέματα των ΦΑΜΠ θα πρέπει να εμπλακούμε για να λυθούν τα προβλήματα Γαλλίας-Γερμανίας. Θα πρέπει κάθε χώρα να προσπαθήσει. Κυρία Μάισνερ, αναφέρατε επίσης την ε, ενοποιημένη πολιτική στις θαλάσσιες ε, μεταφορές. Ο Υπουργό Μεταφορών της Ολλανδίας είναι και Υπουργό Τουρισμού και είμαι υπεύθυνο και για τα λιμάνια και για την ε, ακτοφυλακή. Πάρα πολλές μεγάλο φόρτο εργασίας. Νομίζω λοιπόν ότι πολλά θα γίνουν και στο δικό μας επίπεδο αλλά και στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών και ελπίζω να μπορέσουν να προοδεύσουν. Επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το τέταρτο πακέτο σιδηροδρομικών μεταφορών θέσαν το θέμα η κυρία Μέσνερ και η κυρία Γιάλα Σέντερ. Βεβαίω θέλουμε να προχωρήσουμε μόλις δημοσιευθεί το σχετικό αυτό πακέτο από την Επιτροπή. Για να απαντήσω στην ερώτηση ενός άλλου συναδέλφου σας, δεν μπορούμε να προοδεύσουμε πάρα πολύ γρήγορα σε θέματα τεχνικά και θέματα ασφαλείας διότι είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Uh, και βεβαίω, εάν δεν υπάρχουν ενοποιημένα συστήματα σε θέματα ασφαλή και με διαφορετικά συστήματα, δεν μπορούμε να έχουμε πρόοδο και εξελίξει πολύ γρήγορε. Μιλήσατε επίσης για τα ΔΕΔ στον τομέα των μεταφορών. Εμείς είμαστε ένα νησί και δεν έχουμε τα ίδια προβλήματα που έχουν οι σκανδιναβικές χώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει οι οδηγίες θα πρέπει να γίνονται σωστά και να κάνουμε κάτι τόσο σοβαρό για να διευκολύνουμε τον τομέα. Τώρα όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών εναερίων μεταφορών. Νομίζω ότι ό,τι κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης. Διότι οι, πελάτε, οι, οι, συγγνώμη, πολίτες της Ευρώπης βλέπουν τι πρακτικό μπορεί να κάνει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο στα θέμα του roaming και η μείωση του κόστους της κινητής τηλεφωνίας είναι κάτι το οποίο εκτιμούν οι πολίτες και εμείς θα πρέπει και κάτι παρόμοιο θα πρέπει να κάνουμε και στο θέμα των ε, εναερίων μεταφορών. Τώρα, η ασφάλεια των επιβατών, των ε, επιβατηγών σκαφών, των σκαφών αναψυχής. Μετά από το ατύχημα του Κώστα Κονκόρδη. Επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να περιμένουμε την έκθεση, την έκθεση πρόοδου και θα ζητηθούμε το θέμα αυτό στο Συμβούλιο του Ιουνίου. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχετική νομοθεσία. Και δεν νομίζω θα γίνει κάτι τους επόμενους μήνες. Ο κύριος Κόλιτσεκ ήταν ο πρώτος που ανέφερε τον τουρισμό. Τον ευχαριστώ. Και τα Εμείς δεν έχουμε πολύ σημαντικές ε, εσωτερικές πλωτές μεταφορές όπως η υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης τα θέματα που αφορούν τους οδηγούς των φορτηγών, των, ε, ε τις ώρες ανάπαυσης και εργασίας είναι ένα άλλο θέμα που αναφέρατε. Ε, ο κύριος Βαντάλεν έφερε ένα θέμα που είναι θέμα που αφορά τον ΕΑΣΑ και όχι εμάς. Αλλά η ΕΑΣΑ είναι αυτή που ασχολείται. Αν φτάσει σε εμάς έχει καλώς. Τώρα, τη ΝΕΑ που αναφέρατε. Δεν θέλω να πω τίποτε. Ως Υπουργός Μεταφορών ξέρουμε τι στόλο διαθέτουν, πόσους επιβάτες μεταφέρουν. Μέχρι τώρα σε θέματα ασφαλείας είναι άψογη η Ryanair. Ξέρουμε και πολλές φορές ότι υπάρχουν ε, δημοσιεύματα στον τύπο τα οποία αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων Ryanair που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Αλλά βεβαίως τα θέματα ασφαλείας είναι πολύ σημαντικά. Κυρία Τσικάου αναφέρθηκε στα θέματα της ε, ενοποίησης και εναρμόνισης των αδειών οδήγησης των επαγγελματιών οδηγών και τους ταχογράφους, ο κύριος Κόχ. ότι οι σωστές δομές της μεταφορές θα πρέπει να οδηγούν και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, συμφωνώ και σε ανάπτυξη. Τώρα, όσον αφορά τη συμφωνία ATR, θα προχωρήσουμε. Νομίζω ότι σχεδόν όλα τα θέματα τα κάλυψα. Η ασφάλεια των οδικών μεταφορών επίσης είναι σημαντική. Εμείς πρέπει να σας πω ότι από επικίνδυνη χώρα για τις ε, οδικές μεταφορές είμαστε η τέταρτη, πέμπτη καλύτερη σήμερα, ασφαλέστερη και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας το θέμα αυτό της οδικής ασφάλειας θα το προωθήσουμε όλους ιδιαίτερως. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ήταν εξαιρετικά καρποφόρα αυτή η πρώτη συνάντησή μας στην αρχή της ε, Προεδρίας σας και θα είναι σίγουρα φορτωμένο και πολύπλοκο το πρόγραμμά σας, αλλά συνάμα και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε για την ε, ενεργητικότητά σας επειδή είστε νέος και για τις δεσμεύσεις. Πολύ δυναμικός μας φαίνεστε και μπράβο μας χρειάζονται άνθρωποι σαν και εσάς. Να είστε σίγουρος ότι εμείς θα είμαστε με την Επιτροπή ολόκληρη στο πλευρό σας για να υποστηρίξουμε όλες τις αποφάσεις σας. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ήδη καθυστερήσει. Θα περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, σημαντικό σημείο που έχει να κάνει με την ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού ο κύριος Τσίλερ νομίζω είναι αυτός ο οποίος θα παρουσιάσει την έκθεση αυτή πρωτού ψηφίσουμε γιατί ο κύριος Καμάλα απουσιάζει. Έχετε το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του κυρίου Καμάλ, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Βρίσκεται ακόμα στο τρένο προερχόμενος από το Λονδίνο. Ξέρετε ότι Λίγο χιόνι μπορεί να προκαλέσει πολύ σημαντικές καταστροφές. Θα ήθελα εξ ονόματος του εισηγητή να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν για το νομοθετικό αυτό φάκελο, ιδίως για την επικοδομητική συνεργασία που δείξανε και για τη διάθεση να υποβληθούν συμβαστικές τροπολογίες την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Κατά αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε τρεις συμβαστικές τροπολογίες οι πολιτικές ομάδες κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συνένεση για τα τρία βασικά ζητήματα όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού στις μεταφορές, κυρίως το αεροπορικό πακέτο για το οποίο συνεχίζονται οι πραγματεύσεις, το συνδρομικό πακέτο, καθώς επίσης και τις οδικές μεταφορές για τα βαρέα φορτηγά. Ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορες διστάμενες απόψεις στα τρία αυτά σημεία, ωστόσο όμως ο συγητής θα ήθελε να τονίσει στο υπόλοιπα μέλη ότι πρόκειται για συμβαστικέ τροπολογίες, οι οποίες ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονται στις μεμονωμένες απόψεις που έχουν είτε τα μέλη της Επιτροπής είτε και οι εισηγητέ και συνεισηγητέ. Πάντω, στα πλαίσια ενό επικοδομητικού πνεύματο, ελπίζει ο κύριο ε, Καμάλ ότι θα καταφέρουμε να στείλουμε μια επικοδομητική γνωμοδότηση προ την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσίλε. Ο κύριο Γκρός θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας πω ότι ε, καταφέραμε τελικά στο Στρασβούργο να συνεδριάσουμε οι σκιώδεις συγητές. Και όντως η σε αυτή ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και καταλήξαμε τελικά σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Δεν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με όλες αυτές τις τροπολογίες. Ειλικρινά θα θέλαμε μια πιο κοινωνική προσέγγιση, για να πω το λιγότερο. Για παράδειγμα, όσον αφορά την συμβαστική τροπολογία παριθμών θα θέλαμε κάποια στοιχεία που να έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική. Μια κάποια κοινωνική πτυχή, μια κάποια κοινωνική διάσταση σε αυτή την τροπολογία. Ενδεχομένως η διατύπωση θα μπορούσε να ήταν κάπως πιο στεναρή όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και την προστασία των εν λόγω υπηρεσιών. Ωστόσο, πιστεύω ότι με την παρούσα μορφή του, οι συμβαστικές τροπολογίες θα έχουν τελικά η γενικότερη υποστήριξη στην Επιτροπή μας. Η δική μας πολιτική ομάδα σαφώς υποστηρίζει τον ανταγωνισμό, αλλά όχι πάση θυσία, όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Θεωρούμε ότι η αύξηση του ανταγωνισμού θα επηρεάσει τελικά τα δικαιώματα των εργαζομένων ή και την ποιότητα των υπηρεσιών μεταφορών. Ελπίζω λοιπόν ότι ο εισηγητή και ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα υποστηρίξουν την τροπολογία επαριθμών 33, η οποία αναφέρεται στην συνέχιση του προγράμματος που αναφέρεται στην τροπολογία αυτή και ότι θα υπάρξει μια πιο έντονη υποστήριξη των κοινωνικών πτυχών στις θαλάσσιες μεταφορές και γίνεται επίσης στην τροπολογία αυτή αναφορά στην, στα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν στις ναυτιλιακές εταιρείε προκειμένου να ανανεώσουν το στόλο τους. Ελπίζω ότι θα υποστηρίξετε επίσης την τροπολογία επαριθμών 26 η οποία αναφέρεται στην χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας τεχνολογίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές προκειμένου να έχουμε ένα ενοποιημένο ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης. Ξέρετε ότι τα συστήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζουν πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό. Να καταφέρουμε να ενοποιήσουμε τα συστήματα πλοήγησης θα βελτιώσει τελικά και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πολύ σημαντική για μας είναι επίσης και η τροπολογία παριθμών 4. Η τροπολογία αυτή καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισης της οδηγίας όσον αφορά τις τουριστικές υπηρεσίες και τη σχετική δέσμη μέτρων. Στο πρόγραμμά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει υποσχεθεί να υποβάλει μια σχετική πρόταση, δεν το έχουν κάνει ακόμα αυτό. Θεωρούμε πάντως ότι για την προστασία των τουριστών η νομοθετική αυτή πρόταση είναι όντως πάρα πολύ κρίσιμη. Τέλος, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι η δική μας πολιτική ομάδα προωθεί ανταγωνισμό και ανταγωνιστικότητα, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι οποιαδήποτε μελλοντική πρόταση για απελευθέρωση του τομέα δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της ποιότητας των υπηρεσιών μεταφορών ή εις βάρος των εργαζομένων στον τομέα. Ευχαριστούμε κύριε Μάισνερ εκ το λόγο. Μιλώ εκ μέρους του κυρίου Μπενιάν. Ε, ήταν εδώ αλλά έπρεπε να φύγει. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πω τι είπε σχετικά με τη θέση του σκιώδης συζητητής. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του και τη συνεργασία για αυτή την έκθεση. Η ομάδα μου υποστηρίζει όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες που κατατίθενται σήμερα. Η κυρία Τικάου τη ανέφερε. Η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού είναι μία από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές της Ευρώπης για την πρόθεση του ανταγωνισμού στην Ευρώπη ώστε να παραμείνει καινοτόμος και ανταγωνιστική. Αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει να κάνει με τη δουλειά που χρειάζεται ακόμα να γίνει για να διασφαλίσουμε τον δίκαιο ανταγωνισμό στον τομέα των ε, μεταφορών. Περιμένουμε το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο από την Κομισιόν για να ενισχύσουμε ε, το θέμα αυτό, αλλά και την ασφάλεια στα αεροδρόμια. Επίσης, ε, η Κομισιόν ε, πρέπει να ταυτοποιήσει τους τομείς που έχουν ε, λίγο ή καθόλου ανταγωνισμό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Αυτά από τον σκιώδη εισηγητή μας. Ευχαριστούμε την κυρία Μάισνερ. Τώρα ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ. Σήμερα δεν είναι εδώ εισηγητής, αλλά για πραγματικά για πρώτη φορά Ε, το ότι δεν είναι εδώ δεν οφείλεται σε αυτόν αλλά στους σιδηροδρόμους και πραγματικά υπήρχε ε, τεράστια απογοήτευση για αυτό το θέμα. Υπήρχαν τόσες ε, συμβαστικές τροπολογίες και καμία συζήτηση σε άλλες επιτροπές. Ε, αυτό είναι σύνηθες λένε. Εγώ ποτέ δεν το έζησα εδώ. Ρώτησα αν όντως γίνεται κάτι τέτοιο ε, όταν είναι αυτός ο εισηγητής. Ίσως, ναι. Ε, από αυτή την άποψη λοιπόν έχει δίκιο. Χαίρομαι τέλος πάντων που όπως και να έχει συναντηθήκαμε και για ένα από τους συμβασμούς ε, που διατυπώθηκαν ε, είναι σε δύο μέρη. Θα ψηφίσω υπέρ του ενός και όχι του άλλου. Για το θέμα των μεταφορών αναφέρει τα λόγια του Γιονοχάνες Λουβίνκα που ήταν ένας ήταν γενικός γραμματέας ε, στην κυβέρνηση όταν ε, έγινε η επανένωση της Γερμανίας. Ήταν ε, ε υπουργό Οικονομικών και έλεγε ότι οι μεταφορές είναι η, αγο... η οικονομία των αγορών εκτός δράσης. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλά να κάνουμε. Πραγματικά έχουμε πάει προς την λάθος κατεύθυνση γιατί ως τώρα αυτοί που καταστρέφουν το κλίμα ε, υποστηρίζονται και όλοι οι άλλοι θα, σας, θα βαρεθείτε να μ' ακούτε να λέω τα ίδια ε, δεν ε, προωθούνται και έτσι δεν υπάρχει καθόλου ανταγωνισμός τουλάχιστον έστω ένας κάποιος ανταγωνισμός. Από αυτή την άποψη λοιπόν ως πράσινη είμαστε ικανοποιημένοι αν υπάρχει έστω και λίγος ανταγωνισμός, αν και απέχουμε έτσι φωτός ακόμα από το στόχο μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κράμαρ, ο κύριος Κοϊτσέκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μου φαίνεται ότι οι προτάσεις και οι συμβαστικές τροπολογίες αντικατοπτρίζουν σωστά αυτούς οι οποίοι τις κατέθεσαν τις τροπολογίες. Με ανησυχεί. Στο σημείο 6 το ότι ζητούμε από την Επιτροπή όταν καταθέσει νέες νομοθετικές δέσμες με τους λιμένες να εμπνευστεί από την ε, εμπειρία κάποιων κρατών για την ιδιωτικοποίηση και να ακούσει τι έχει να πει η αγορά, ώστε να δημιουργηθεί ένα ανοιχτό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τώρα όσον αφορά τις εναέριες μεταφορές, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα υποχρεώσουμε τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες πέραν του Ατλαντικού να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε. Η κοινωνική διάσταση και καλύτερες συνθήκες εργασίας για να έχουν καλύτερο ανταγωνισμό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ισχύει σε όλους τους τομείς των μεταφορών. Κυρίως για τις οδικές μεταφορές είναι χαόδης η κατάσταση όσον αφορά τι συνθήκε εργασία. Για τα μεγάλα φορτηγά Όλοι ενδιαφέρονται. Όταν έχουμε όμως μικρότερα, μικρότερα από 3,5 τόνους, είναι καταστροφική η κατάσταση που επικρατεί. Και επίσης, όσον αφορά την ε, υπηρεσία σε εδάφους, τα πράγματα επίσης δεν είναι σωστά και φοβούμε ότι υπάρχει κίνδυνος για τις κοινωνικές συνθήκες και για το κοινωνικό κράτος το οποίο θα πρέπει να έχουμε δεδομένο ότι αυτό πρέπει να αποτελεί μια από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω αμέσως ε, ε, να πω ότι πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εκ, τους, εκ μέρους του συναδέλφου. Υπάρχουν πολλά προβλήματα μεταφορών. Νομίζω ότι με αυτή την ε, έκθεση έχουμε μία ετήσια άσκηση, ας πούμε, που ε, πραγματικά οδήγησε σε συμβιβασμό μεταξύ των ε, συντονιστών. Θεωρώ ότι δεν συμφωνώ με τις ε, θέσεις της Κομισιόν για τη φορολογία στους σιδηροδρόμους. Εδώ και πάνω από δύο χρόνια η Κομισιόν δεν έχει κάποια συγκεκριμένη θέση σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που εισάγουν φόρους και αυτό είναι κατά του ελεύθερου ανταγωνισμού και των συνδεδόμων γενικότερα. Συμφωνώ και με την πρόθεση επιπλέον κοινωνικών στάνταρ διαπιστώνω ότι Υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις για τον ανταγωνισμό στη δέσμη μέτρων, όμως ε, ο ανταγωνισμός χωρίς δίκαιους κανόνες και κοινωνικά στάνταρ δεν είναι δίκαιος ανταγωνισμός. Και για το κείμενο από πέρσι να πω ότι είναι καλύτερο αυτό και θα πρέπει να γίνουν δεκτέ οι συμβιβασμοί. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ρικέ. C'était Πολύ ωραία το οργανώσαμε το θέμα. Θα ήθελα να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω την εργασία τους και τον εισηγητή και γιατί εγώ προσωπικά θα ήθελα να υποβάλω ένα αίτημα. Μια στιγμή γιατί έχω χαθεί εδώ στα χαρτιά μου επειδή μπήκε ο Μπράιαν στην αίθουσα. Θα ήθελα να ζητήσω οι τροπολογίες μου μια στιγμή. Λοιπόν, η τροπολογία 37 να υπερψηφιστεί, διότι πιστεύω ότι δεν συμπεριλαμβάνει τη συμβαστική τροπολογία 3. Το ίδιο με τη 43 που δεν είναι συμβαστική τροπολογία 4. Ε, Άκουσα προηγουμένως την κυρία Τσικάου να λέει ότι η κοινωνική διάσταση εδώ δεν τονίζεται ιδιαιτέρως, ε, συμπεριλαμβάνεται στις δικές μου τροπολογίες. Οι 37 λοιπόν και 43 τροπολογίες μου δεν καλύπτονται. Δεν θα ήθελα να εξαφανιστούν. Ζητώ λοιπόν να ψηφιστούν. Το ζητώ αυτό διότι είναι δικαίωμά μου να επιμείνω. Παρακαλώ λοιπόν να ψηφίσουμε αυτές τις τροπολογίες 37 και 43. Ο Μάικλ, θέλεις να επανέλθεις σε κάτι? I had forgotten something. Ah, ja, ich habe noch eins vergessen. Wir haben ja einen Änderungsantrag Nummer 30. Έχουμε την τροπολογία 30, το ξέχασε. Και εκεί ζητούμε από την Κομισιόν ένα νέο νομοθετικό πακέτο. Και αυτό είναι λίγο σκληρό θα έλεγα. Ε, αύριο θα κάνουμε μια προφορική τροπολογία και θα σκεφτείτε αν είστε υπέρ ή κατά. Εγώ χαίρομαι να, θα χαρώ να είστε υπέρ φυσικά. Η Κομισιόν όταν ε, προβάλλει νέα μέτρα για τα λιμάνια, όχι, όχι νέο νομοθετικό ε, πακέτο, για να μάθουμε από τους επαγγελματίες και την πρακτική εμπειρία έτσι ώστε να έχουμε μία αποτελεσματική προσέγγιση που θα προσανατολίζεται στι ανάγκε τη αγοράς αλλά και σε ικανοποιητικές συνθήκε εργασίας. Άρα προχωράμε σε επέκταση του πεδίου, όχι σε νέα νομοθετική πρόταση. Η κυρία Πρόμψ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα σχολιάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες αυτές καθεαυτές. Θέλουμε να σας δώσουμε απάντηση στην ερώτηση που παρουσιάστηκε στην συνάντηση της Επιτροπής ε, το Δεκέμβρη. Ο κύριος Σίμψον μίλησε για το θέμα ε, του Manchester Route και το θέμα της συμπροευρίας μεταξύ των Brussels Airlines και της Flybe. Αυτή τη στιγμή διαρευνούνται ε, δύο περιπτώσεις για να δούμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα του code sharing. Έχοντας ε, δει την κατάσταση στην διαδρομή Βρυξέλλες-Μάντσεστερ φαίνεται ότι είναι το wet lease και όχι code sharing που ισχύει. Το wet lease σημαίνει ότι μία αεροπορική εταιρεία δίνει ένα ελεύθερο ε, ε, αεροσκάφο σε μια άλλη με αποζημίωση. Χωρίς ε, τους πιλότους, χωρίς το προσωπικό και χωρίς και τα πιστοποιητικά. Γι' αυτό η Brussels Airlines θεωρεί ότι η άλλη εταιρεία είναι αυτή που λειτουργεί την πτήση. Οι πτήσεις όμως αυτές ε, δεν πολλούνται ως πτήσεις Flybe και δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα της Flybe. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα. Γι' αυτό η κατάσταση δεν έχει να κάνει με τη συνεχή έρευνα για το code sharing. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Τζίλε που Σας ευχαριστώ πολύ. Θα διαβιβάσω όλες αυτές τις πληροφορίες στον κύριο Καμάλ. Μου κάνει εντύπωση το ότι γίνανε τόσο πολλές συναφορές από όλες τις πολιτικές ομάδες στην κοινωνική διάσταση. Ξέρετε ότι τα κοινωνικά αυτά ζητήματα είναι προβληματικά και δύσκολα από πολιτικής πλευράς. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να τα εντάξουμε σε μια καλή πολιτική ανταγωνισμού. πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία είναι αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Ντομινίκ, σε ευχαριστώ πολύ που με αντικατέστησες κατά τη διάρκεια της καθυστερισμένης μου πτήσης από το Μάντζεστερ. 7,5 ώρες καθυστέρηση. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, υπηρεσίες εδάφου στεροδρόμια της Ένωσης και κατάργηση οδηγίας 1667. Ο κύριος Τζαζάντα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Δεκέμβριο Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που κάναμε στην Ολομέλεια, αποφασίσαμε να αποστείλουμε το κείμενο αυτό πίσω στην Επιτροπή Μεταφορών και οι στονιστές μου δώσαν εντολή προκειμένου να καταφέρουν να συνεχίσουν να επεξεργάζομαι την συμβαστική αυτή λύση για τις υπηρεσίες εδάφους στα αεροδρόμια. Στόχος μου είναι να καταφέρω να εξασφαλίσω μία πλειοψηφία προκειμένου να εγκριθεί το κείμενο αυτό στην Επιτροπή μας. Γι' αυτό το λόγο διοργάνωσα δύο συναντήσεις με τους κοιόδες ηγητές και στη συνέχεια επέβαλα ένα θεωρημένο κείμενο της λεγόμενης συμβαστικής Α και προτίμασα και ένα νέο συμβαστικό κείμενο I. Οι βασικές αλλαγές έχουν να κάνουν ε, με το κατόφλι από τα 5 που πήγε στα 15 εκατομμύρια και έχει επεκταθεί η περίοδος εφαρμογής από ένα, χρόνια, από ένα έτος σε τρία χρόνια και έχουμε ουσιαστικά διπλασιάσει το χρόνο που προβλεπόταν στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προκειμένου να καταφέρουμε να αποκριθούμε στα των σοσιαλιστών, θα κινδύνευα ουσιαστικά να χάσω την υποστήριξη των συναδέλφων εκείνων που με είχαν υποστηρίξει από την αρχή και που θέλαν την απελευθέρωση των υπηρεσιών εδάφου. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Δυστυχώ τα περισσότερα αιτήματα των σαλιστών είχαν να κάνουν με αυτό το συγκεκριμένο τμήμα του κειμένου, το οποίο ουσιαστικά δεν υπάγεται στη δική μου την αρμοδιότητα, το οποίο εγώ δεν μπορώ συγητή να τροποποιήσω. Ουσιαστικά αναφέρομαι στην γνωμοδότηση επιτροπή απασχόληση σύμφωνα με τον κανόνα 50. Οι σοσιαλιστές ουσιαστικά θέλανε να υπάρχουν ε, οι υποχρεωτικές μεταφορές ε, προσωπικού για όλες τις κατηγορίες, ε, ενώ εδώ πέρα η Πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει μόνο μία εθελούσια τέτοια μεταφορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε μία κοινή θέση με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είχαμε μείνει στη θέση των σοσιαλιστών. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε μία συμφωνία με τους σοσιαλιστές και με τον κύριο Μάν που εκπροσωπεί την Επιτροπή Απασχόλησης. Η συμφωνία ενδεχομένω αυτή να είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Γι' αυτό το λόγο σας υποβάλλω δύο εναλλακτικέ. Πρώτη, να γίνει μια κοινή συνεδρίαση όλων των σχεδόν εισηγητών της Επιτροπής Μεταφορών αλλά και της Επιτροπής Απασχόλησης, προκειμένου να συνεργαστούμε από κοινού για μια λύση η οποία θα ικανοποιήσει όλες τις πλευρές. Νομίζω ότι αυτό είναι ο μόνο τρόπο που έχουμε προκειμένου να ξεπεράσουμε τι δυσκολίε που έχουμε μπροστά μα. Και αυτό μου προτείνει άλλωστε και η γραμματεία. Το αδύναμο σημείο όμω τη λύση αυτή είναι ότι οι συντονιστέ από την Επιτροπή Απασχόληση αποφάσισαν στη δική του συνεδρίαση την Πέμπτη να μην ανοίξουν εκ νέου το κείμενο αυτό. Και δεν μα είχε δοθεί καμία διασφάλιση ότι το νέο κείμενο θα έχει την υποστήριξη όλων. Δεύτερη εναλλακτική τώρα την οποία εγώ βρίσκω πολύ δύσκολη, αλλά θα αποτελέσει ουσιαστικά μια ίστατη προσπάθεια για να πετύχουμε ένα κάποιο συμβασμό. Σας προτείνω ο συμβασμός υπαριθμών α να λέει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω απελευθέρωση των υπηρεσιών εδάφου θα εναπόκειται πλέον σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αποκλειστικά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για τα αεροδρόμια άνω των 2 εκατομμυρίων επιβατών και πάνω από 50.000 τόνους φορτίου, ένα οποιοδήποτε κράτος μέλος, ένα δεδομένο κράτος μέλος, δεν θα μπορέσει να περιορίσει τους φορείς παροχής υπηρεσιών εδάφους σε λιγότερους από δύο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τη λύση αυτή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς με την πρόταση αυτή ή με μία από τις δύο εναλλακτικέ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λόγος, ότι αξίζει πραγματικά να προωθήσουμε περισσότερο το κείμενο αυτό και να το επεξεργαστούμε περισσότερο. Σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, οι επιβάτες γνωρίζουν πάρα πολλά προβλήματα, είτε έχει απελευθερωθεί η αγορά είτε όχι. Βλέπω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο ή στη Φραγκφούρτη και βλέπω ότι τελικά το τίμημα το πληρώνουν οι ίδιοι οι επιβάτες, οι οποίοι για έξι ώρε και παραπάνω τελικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αφήνονται στο έρμεο τελικά τη κακοκαιρία χωρί να του δίδεται καμία απολύτως πληροφορία. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί τελικά δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός ο οποίος θα επέτρεπε σε έναν φορέα εκμετάλλευση των αερολιμένων να ασκήσει πίεση προκειμένου να ανοίξουν να δοθούν, με συγχωρείτε, κάποιες πληροφορίες. Θεωρώ λοιπόν ότι οι προτάσει οι οποίε περιλαμβάνονται κυρίω στο παράρτημα τη πρόταση κανονισμού μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν πολύ περισσότερο από μια νέα νομοθετική πρόταση μετά από 10 χρόνια. Ξέρετε ότι δεν μπορούν οι επιβάτε να περιμένουν τόσο πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση και για τα 27 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε μια ομοιόμορφη προσέγγιση πανευρωπαϊκώ. Θεωρώ ότι είμαι πραγματικά υπεύθυνο για την πρόταση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν σας προτείνω να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές ομάδες βάσει των προϋποθέσεων που σας πρότεινα. Οποιαδήποτε περαιτέρω απελευθέρωση θα είναι απόφαση μεμονωμένων κρατών μελών. Αν τελικά συμφωνήσουμε με την πρόταση αυτή, μπορούμε να ψηφίσουμε εκ νέου στην Επιτροπή μας το Φεβρουάριο και να πάει η πρόταση αυτή στην Ολομέλεια τον Μάρτιο-τον Απρίλιο. Με τη δική σας λοιπόν σύμφωνη γνώμη θα μπορούσαμε βάσει του κανόνα 56 να υποβάλουμε την πρόταση αυτή και να πούμε ότι θα ψηφίσουμε το αργότερο στις 12 Φεβρουαρίου. Πρόεδρος, μπορούν οι σκιώδεις να πάρουν τώρα το λόγο, αλλά να μιλήσουν για δύο λεπτά μόνο ο κύριος Φλέκενστάιν πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω ότι είπαμε ότι μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι συμβεβασμοί. Έξι είναι τα σημεία που αναφέραμε. Ο εισηγητής ανέφερε ποια είναι τα σημαντικά. Αυτή τη βδομάδα η ΕΜΠΛ ε, συνεδριάζει και θα συζητηθεί το θέμα έτσι ώστε να βγει το όλο πακέτο και αυτό το περιμένουμε και μετά θα δούμε τι θα βγει από αυτό. Αυτό που δεν θεωρούμε σωστό σε καμία περίπτωση είναι να αποφασίσουμε κάτι που μετά θα είχε νόημα μόνο αν από την άλλη πλευρά υπήρχε και αντίστοιχη ε, πρόοδος. Η πρόταση του εισηγητή σε επίπεδο ε, ορίων Μόνοι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και θεωρώ, α, πρέπει να το συζητήσουμε και στην ομάδα μας βέβαια, ότι δεν θα θέλαμε να ψηφίσουμε κάτι που στο τέλος θα το αρνηθεί η Ολομέλεια γιατί δεν ταιριάζει με, το, με την όλη εικόνα. Είτε πρόκειται για περαιτέρω απελευθεροποίηση, είτε όπως και να το πούμε, πάντοτε υπάρχουν ε, οι κοινωνικοί μοχλοί που πρέπει και αυτοί να ρυθμίζονται κατάλληλα. Δεν είναι μεγάλη καταστροφή που διαγράφεται αυτή η τροπολογία. Από την άλλη έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν και ο εισηγητής θα μπορούσαν να τα μειώσουν στην πρόταση η Φραγκφούρτη θα, θα έπρεπε να έχει το 1 τρίτο και αυτό θα μας ε, ενδιέφερε όλους νομίζω. Ευχαριστώ Κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ. Καταρχάς ε, ευχαριστώ τον εισηγητή. Κρίμα που κουράζεται Τόσο, εμείς ε, οι φιλελεύθεροι έχουμε από τη μία υποστηρίξει την πρότασή του γιατί η βασική ιδέα της απελευθερώσης ε, στηρίζεται, όμως έχουμε και κάποιες αμφιβολίες έχουν ως εξής. Καταρχάς, θεωρούμε, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, ασχολούμαστε με το θέμα αυτό ε, για λίγα αεροδρόμια τελικά. Ταυτόχρονα όμως ε, εισάγουμε και αλλαγές μέσα από αυτά που ε, υποστηρίζει η Επιτροπή ε, Απασχόλησης για παράδειγμα που αγγίζουν όλα τα αεροδρόμια. Δεν είναι και πολύ σωστό αυτό, πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν. Δεύτερον, θέλουμε ένα ενιαίους διαγωνισμούς με τις ίδιες αρχές έτσι ώστε να φροντίζουν τον ανταγωνισμό. Τώρα αν είναι αναγκαίο σε όλες τις χώρες να έχουμε μια αρχή αδειοδότησης ε, με τις ίδιες αρχές, ε, με τη, που θα βασίζεται στις ίδιες αρχές, δεν ξέρω. Αυτό ίσως να οδηγεί σε μεγάλη γραφειοκρατία και ακριβώς σε αυτό το σημείο τα μικρά αεροδρόμια θα έχουν μειονέκτημα. Πάμε ένα βήμα πιο πέρα δηλαδή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι από τη μία πλευρά θέλουμε ίδιους όρους ανταγωνισμού, απ' την άλλη όμως λέμε ότι η Ευρώπη πάρα πολύ εμπλέκεται στις υποθέσεις των κρατών μελών που θα μπορούσαν να λύσουν μόνα τους. Και εδώ είναι ένα τέτοιο θέμα. Ουσιαστικά ε, ζητείται από τα κράτη-μέλη να γίνονται περαιτέρω περικοπές εμείς ε, λέμε τουλάχιστον δύο, οι άλλοι ίσως ε, αποφασίζουν μόνοι τους αν θέλουν παραπάνω, όμως τελικά ίσως πάμε ανάποδα. Βλέπω τον κίνδυνο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πει ότι απελευθερώνουμε τις ε, υπηρεσίες εδάφους και de facto δεν γίνεται τίποτα. Τότε πραγματικά ε, οδηγούμαστε σε μια τρελή κατάσταση, μπερδεύουμε τους πολίτες. Και ένα τελευταίο σημείο. Αν, μπορούμε να υποσχε... Αν υποσχεθούμε πολλά, το είπε πριν και ο προλαλής σας, ο Τόμας Μαν και εδώ η, η αν μπορούν η δική μας Επιτροπή και Επιτροπή ε, ε, ε να έρθουν, να συνέλθουν και να ε, μιλήσουν και να συζητήσουν, ίσως θα μπορούσα εγώ να συμφωνήσω. Η κυρία Λίχτενμπεργκερ, να πω εξ αρχής ως επιφύλαξη ότι έχουμε ε, μεγάλη σπατάλη λόγω του δύο στριών 3 operators σε λίγα ε, αεροδρόμια στην Ευρώπη και για ένα διάστημα μεταβατικό. Οι πολίτες δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και όπως είπε και ο συνάδελφος Κλίντς, διαψεύδουμε προσδοκίες. Μιλάμε για απελευθέρωση, αλλά τελικά είναι περιορισμένη απελευθέρωση. Από τη δική μου πλευρά, λοιπόν, όλο αυτό το θέμα είναι δύσκολο στην επεξεργασία του, γιατί πηγαίνει προς μια κατεύθυνση και όταν εδώ στην Επιτροπή βάζουμε κάποια φρένα και δεν προχωρά το θέμα, τότε γίνεται πολύ πολύπλοκο. Έτσι λοιπόν το πιο έξυπνο θα ήταν η Κομισιόν να έπαιρνε πίσω αυτό το θέμα και να το ξανακοίταζε γιατί είναι δύσκολο να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την πρόταση με τον τρόπο που γίνεται τώρα. Έχουμε τέλος πάντων ένα νομοσχέδιο που στην ουσία ισχύει για λίγα αεροδρόμια. Το να έχουμε ε, ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, ε, εντάξει είναι σωστό, όμως ε, σε, κάποιες, σε κάποιους τομείς έχουμε ολιγοπόλια και πολλές φορές οδηγούμε σε αντιπαραθέσεις μεταξύ ενός μικρού ολιγοπολίου. Αυτά για τον ανταγωνισμό. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά φέρνει κέρδος στους επιβάτες. Εγώ πραγματικά δυστυχώς ταξιδεύω πολύ και ως ε, επιβάτης ε, δεν μπορώ να διαπιστώσω κάποια πλεονεκτήματα αν είναι απελευθερωμένα ή όχι τα αεροδρόμια. Τώρα για τον τρόπο εργασίας και το πώς θα πάμε παραπάνω. Το αποφασιστικό είναι πώς θα αποφασίσει η Επιτροπή Απασχόλησης, γιατί αν έχουμε διαφορετικές αποφάσεις στις διάφορες επιτροπές, με αυτόν τον κανόνα 56-57 δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Πώς θα το κάνουμε. Πρότειναν οι σοσιαλδημοκράτες συμβεβασμό έναντι του ΕΛΚ και από αυτού πρόκειται τελικά. Αλλά αυτό ισχύει στη μία επιτροπή και στην άλλη που ασχολείται με το θέμα όχι. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια πολύπλοκη κατάσταση. Αν λοιπόν πρόκειτο για ένα θέμα που θα κινούσε τον κόσμο και τουλάχιστον την Ευρώπη τόσο σημαντικό δηλαδή, καλό θα ήταν να το κάνουμε έτσι και να κάτσουμε ένας με τον άλλον, να συζητήσουμε και να δούμε τι περιθώρια συνεργασίας έχουμε. Όμως το καλύτερο θα ήταν να ζητήσουμε από την Κομισιόν να αποσύρει την πρόταση, να κάνουν μια νέα πρόταση με βάση τα όσα άκουσαν, με πιο απλούς όρους. Θα πάμε πιο πέρα από ότι αν έχουμε ένα πολύπλοκο νομοθέτημα και πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ προβληματικό έτσι όπως έχει το πράγμα. Ευχαριστώ. Έχω πάρα πολλούς που θέλουν να μιλήσουν, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ο κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Στην Ολομέλεια η ομάδα μου είχε πει ότι θα πρέπει το θέμα αυτό να επανέλθει στην Επιτροπή. Δυστυχώς όμως δεν βλέπω να υπάρχει πρόοδος. Απλώς διαπιστώνω ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΕΛΚ και Σοσιαλιστών για να παραταθούν οι προθεσμίες ώστε να μην έχουμε μία πάρα πολύ ε, πακτή γραφειοκρατία, τα δικαιώματα των υπαλλήλων να είναι καλύτερα από αυτά των επιβατών και η Επιτροπή είναι έτοιμη να επανέλθει σε διάφορα θέματα τα οποία είχε εκθέσει. Εκτιμώ τις προσπάθειες του εισηγητού που προσπαθεί να βρει λύσει που ικανοποιούν του πάντες, αλλά την εντύπωση ότι δεν θα το κατορθώσουμε τελικά. Η ιδέα όλο το πακέτο να γυρίσει πίσω στα κράτη-μέλη για νέες προτάσεις μου δημιουργεί ερωτηματικά, διότι θα παραμείνουμε σε αυτό το αδιέξοδο. Φοβούμαι λοιπόν ότι η ομάδα μου θα αντιταχθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι κατ' εξαίρεση συμφωνώ με τον προλαλήσαντα και θα ήθελα να αναφέρω τους κανόνες 56-57 που απαιτούν να λάβουμε υπόψη της τροπολογίας. Δηλαδή, να έχουμε μια νέα πρόταση και να εξετάσουμε τις τροπολογίες βάσει του 56-57. Διότι αν υπάρξει σε επίπεδο ολομέλειας δύο φορές άρνηση και αν επανέλθει και πάλι για δεύτερη φορά στην ε, Επιτροπή μας θα χρειαζόμαστε μια νέα πρόταση για να βρεθεί μια κάποια λύση να προχωρήσουμε. Έτσι, το έγγραφο αυτό, έτσι ως έχει, πρέπει να πω την άχρηστο, δεν προσφέρει τίποτε. Λοιπόν, έχω ακόμη τρεις υποψήφιους ομιλητές. Τρεις συντονιστές. Θα πρέπει να έχουμε τελειώσει, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε και να τελειώσουμε γρήγορα να αρχίσουμε και την συνεδρία συντονιστών. Ο κύριος Γκρός, πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε στο ΕΛΚ είχαμε συμφωνήσουμε ε, Είχαμε συμφωνήσει ότι θα προσπαθήσουμε να δούμε αν έχουμε προστιθέμενη ε, αξία. Ο συνάδελφος Σασάγα είπε ότι είναι έτοιμος, έδειξε ότι είναι έτοιμος ε, για συμβιβασμούς. Είναι ενδιαφέρον ότι από τα σχόλια των συναδέλφων βλέπουμε τώρα ότι στην αρχή έβλεπαν τα πράγματα ότι δεν είναι τόσο κοινωνικά, τώρα τα βλέπουν ότι είναι υπερβολικά κοινωνικά. Ε, μετά μιλήσανε για στρέβλους του ανταγωνισμού. Έχω το αίσθημα ότι το σημαντικό είναι να αποσυρθεί το ντοσιέ και παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τα πράγματα. Θα χρησιμοποιήσουμε όμως την ευκαιρία να βελτιώσουμε λίγο τα πράγματα. Δεν είναι απλό έτσι να δώσουμε πίσω τον τοσχέ στην Κομισιόν, γιατί θεωρούμε ότι η τωρινή κατάσταση με τις υπηρεσίες ε, εδάφους ε, μπορεί να βελτιωθεί και για τους επιβάτες και για τους εργαζομένους. Θα ήθελα να πω ότι παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι λίγο υπερβολικό το θέμα, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση και τους εργαζομένους, να έχουμε βελτίωση των κανόνων της αγοράς, έτσι ώστε τελικά οι επιβάτες να έχουν κατάλληλες υπηρεσίες. Αυτός είναι ο στόχος. Αν δεν ε, επιτευχθεί, θα βγει και το άλλο από την ε, συζήτηση και καλό θα ήταν να διερευνήσουμε ε, τις δυνατότητες με τους σχεώδεις από τις δύο επιτροπές και μετά να έρθει η συζήτηση ξανά εδώ, ώστε να μην μακρο, μακρηγορήσουμε. Ευχαριστώ και για το χειροκρότημα. Αν πω ότι ήταν από τον Μιχαήλ, μπορεί να μην χαρίσει και τόσο. Πρώτα ο κύριος και μετά εσύ, Μάικλ. Κύριε Πρόεδρε, αρχίζοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να προχωρήσουμε προς την σωστή κατεύθυνση. Εμείς δεν θέλουμε να υποχρεώσουμε τα κρατη να έχουν τουλάχιστον τρεις φορείς παροχής υπηρεσιών. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αλλά εντάξει, ας εξεταστεί το όλο θέμα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανοποιητικό το status quo. Και η οριστική απόρριψη πρόταση θα σημαίνει ότι παραμένουμε στην κατάσταση ως έχει. Πράγμα που δεν είναι πολύ ικανοποιητικό. Άρα είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε το όλο θέμα και να δούμε εάν μπορούμε ενδεχομένως να καταλήξουμε σε συμφωνία, να παραταθεί, να παρατώθουν οι προθεσμίες, αλλά κυρίως να βελτιωθεί η όλη κατάσταση, κυρίως ε, για όλο το πακέτο το οποίο χειρίζονται οι συνάδελφοι της Επιτροπής Απασχόλησης. Η ποιότητα είναι σημαντική, η κατάρτιση είναι σημαντική, οι συλλογικές συμβάσεις οι συνθήκες εργασίες πρέπει να είναι οι ίδιες για όλους, η πρόσληψη του, και η όρη πρόσληψης του προσωπικού, οι συμβάσεις, όλα αυτά τα θέματα. Προτείνω λοιπόν, όπως πρότεινε και ο εισηγητής, να κάνουμε μία από κοινού συνάντηση με τους ε, εισηγητές, και τους χιλιάδες εισηγητές της Επιτροπής με την Επιτροπή Απασχόληση. Και οι συντονιστέ, αν το επιθυμούν, μπορούν να παραστούν και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μια συμφωνία επί του συνόλου και να ψηφίσουμε στην Επιτροπή, μετα... στην Επιτροπή Μεταφορών όλα τα προβληματικά κομμάτια. Βεβαίω θα πρέπει να ξανανοίξουμε γενικά τη συζήτηση, αλλά προφανώς στην Επιτροπή Απασχόλησης θα μπορούσαν να δεχθούν κάποιες συμβαστικές τροπολογίες, τις οποίες θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε στην Ολομέλεια. Και τα θέματα που χειριζόμαστε εμείς δεν θα πρέπει να τα βλέπουμε στα θέματα τα οποία χειρίζεται μόνον η άλλη Επιτροπή. Συμπερασματικά λοιπόν, θα ήθελα να συστήσω στον εισηγητή να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. να γίνει συνεδρίαση των Επιτροπών Μεταφορών και Απασχόλησης και να δούμε αν επί του συνόλου μπορούμε να προχωρήσουμε. Και ελπίζω ότι θα επιχειρεί. Μην έχουμε. Τουλάχιστον θα το έχουμε προσπαθήσει. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από μερικές εβδομάδες αποφασίσαμε να, επιστρέψει η πρόταση αυτή στην Επιτροπή Μεταφορών και ξέρουμε ότι δίστανται οι απόψεις στις πολιτικές ομάδες. Ορισμένοι πιστεύουν ότι δεν προωθείται πάρα πολύ η πτυχή της απασχόλησης. Άλλοι θεωρούν ότι ενδυναμώνται ιδιαίτερα τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι προχωράμε πάρα πολύ με την απελευθέρωση. Άλλοι πάλι ότι δεν προχωράμε αρκετά. Πρέπει όμως να προσεγγίσουμε την πρόταση αυτή συνολικά, σφαιρικά. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να βρούμε μία λύση. Να δούμε δηλαδή πώς θα καταφέρουμε να προωθήσουμε αυτή τη δέσμη μέτρων περαιτέρω, και τι επεξεργασία μπορούμε να τις επιφυλάξουμε για το μέλλον. Νομίζω ότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μια πάρα πολύ καλή βάση. Υποβλήθησαν πολλέ τροπολογίε από τη δεξιά και την αριστερά. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να καταλήξουμε στην παρούσα φάση στις συμβαστικές τροπολογίες. Ενδεχομένως λοιπόν να μα καλύπτει αυτή τη στιγμή η αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής όσον αφορά την απλούστευση, όσον αφορά τη διαφάνεια. Υπάρχουν τα εξή σημαντικά ζητήματα. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εδάφου δεν είναι καλή. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε μία αύξηση της ποιότητας αυτής, να υπάρχουν δηλαδή πιο αυστηρά πρότυπα. Από την άλλη θα πρέπει να εργαστούμε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ε, δεν θα αποτελέσουμε εμεί εμπόδιο για τους επιχειρηματίες. Και συμφωνούσα αστικά με τον κύριο Γκρός. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες συγκεκριμένε λύσεις επιτέλους. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πιο ποιοτικέ υπηρεσίες εδάφους για τους επιβάτες. Η δική μου πολιτική ομάδα θεωρεί ότι ο στόχος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν θέλουμε όμως να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε πρόταση προκειμένου να καταλήξουμε τελικά σε μεγαλύτερη απελευθέρωση του κλάδου. και να εγκρίνουμε τελικά πάρα πολλές ε, νέες κοινωνικές διατάξεις, χωρίς όμως να είναι τελικά το μοντέλο αποτελεσματικό. Τώρα, αν ε, αυτό ε, έχει να κάνει με δύο ή τρία αεροδρόμια και αν θα είναι σχετικό σε 10-15 χρόνια, αυτό είναι το θέμα. Όλοι συζητούμε, βρήκαμε μια θέση με μικρή πλειοψηφία, όμως στην Ολομέλεια ήταν όλοι κατά. Άρα οι ίδιοι συνεχίζουμε μια δεύτερη συζήτηση για το ίδιο θέμα. Δεν είμαστε εμεί αυτοί που θα βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά από την, για λογαριασμό της Κομισιόν που απέτυχε στην πρότασή της. Δεν προχωρεί η πρόταση και αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε. Αυτοί πρέπει να δουν αν θα πάρουν πίσω την πρόταση ή αν θα φέρουν καινούρια με αλλαγές. Είναι δική τους δουλειά αυτή. Από αυτούς πρέπει να το ζητήσουμε μια ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία για τρία μόνο αεροδρόμια είναι τρελό. Έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν. Ξέρω 10, 20, 30 βασικά θέματα με τα οποία θα μπορούσε να ασχοληθεί η Κομισιόν και τελικά ασχολείται με τη Φραγκφούρτη, τη Βιέννη, το Βερολίνο. Άρα εμείς πρέπει να σταματήσουμε με αυτό το θέμα. Η Κομισιόν να δει αν έμαθε το μάθημά τη, να δει αν θα φέρει καινούρια πρόταση, αλλά δεν είναι δική μα δουλειά αυτή. Εμεί γελιοποιούμαστε, έχουμε μια θέση, την ψηφίσαμε. Με μικρή πλειοψηφία στην ε, Επιτροπή, μεγάλη στην Ολομέλεια, η Κομισιόν είναι αυτή που θα πρέπει να αποφασίσει και όχι εμείς. Ο κύριος Γκάλερ. Ναι, ευχαριστώ. Θεωρώ ότι αυτό που πρότεινε ο εισηγητής πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί ε, συνάδελφοι και όχι όλοι, ε, θεωρούν ότι δεν υπάρχει άμεσος ε, δασμός μεταξύ της ποιότητας και του αριθμού. Υπάρχουν αεροδρόμια με λίγους operators που έχουν καλή ποιότητα και μεγάλα με πολλούς που δεν έχουν καλή ποιότητα. Τέλος πάντων, η βελτίωση της ποιότητας μέσω περισσότερων φορέων λειτουργίας ε, δεν ε, είναι αυτονόητο ό,τι συμβαίνει. Για τους σοσιαλδημοκράτες ε, υπόθηκε ξεκάθαρα όταν υπάρχει υποχρέωση για απελευθέρωση θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και σε κοινωνικό επίπεδο. Για μένα όμως είναι ανάποδο το θέμα. Αν δεν υπάρχει υποχρέωση απελευθέρωσης το αφήνουμε δηλαδή στα κράτη-μέλη, τότε καλό θα ήταν να γυρίσουμε και τον μοχλό των κοινωνικών υποθέσεων. Θεωρώ ότι <coughs> δεν πρέπει να κάνουμε κοινωνική πολιτική μέσα από την πολιτική μεταφορών. Η κοινωνική πολιτική και η πολιτική των μισθών πρέπει να γίνεται από τα κράτη-μέλη και όχι μέσα από τις μεταφορές. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι καλή η πρόταση του εισηγητή να αφήσουμε τον τρίτο φορέα στην ε, διακριτική των κρατών μελών και ε, σύμφωνα και με τις ε, ε, προτάσεις της Επιτροπής Αποσχόλησης. αν δεν υπάρχει υποχρέωση απελευθέρωσης, τότε καταπίπτει και αυτό. Ε, παρακαλώ, μέσω του Προέδρου να γίνονται συζητήσεις. κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παναρχόμαστε στην κατάσταση στην Ομοσπονδιακή Γερμανία με όλα αυτά που λέμε. Ευχαριστώ τον ε, συνάδελφο Τσαζάντα για την πρότασή του. Νομίζω ότι εξ αρχής αυτό το θέμα δεν αντιμετώπιζε ε, επαρκώς το θέμα της ε, διαφορετικότητας των αεροδρομίων και των κρατών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πιο στενά το θέμα της επικουρικότητας και να υπάρχει ένα συμβασμό σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι η επικορικότητα ε, πρέπει να συνδέεται και με τη βελτίωση της ποιότητας, το είπε και ο συνάδελφος πριν. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή. Αν ε, στείλουμε το θέμα πίσω στην Κομισιόν, σίγουρα η Κομισιόν ε, δεν θα μπορέσει να καταθέσει νέα πρόταση γρήγορα και σωστά και γι' αυτό καλό θα ήταν να προωθήσουμε το θέμα της βελτίωσης της ποιότητας και των κοινωνικών, της κοινωνικής διάστασης στην έκθεσή μας και σε συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια συνεκτική έκθεση ε, ώστε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πριν φέρω τον εισηγητή να μιλήσει, να σας θυμίσω ως πρόεδρος για τη διαδικασία για το θέμα των υπηρεσιών εδάφους. Αναφέρθηκε πριν κάποιος σε αυτό, είπατε ότι ίσως να υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει εκ μέρους σας να αναφέρω γραπτός ότι να, τι γίνεται πριν τη 12η Φεβρουαρίου. Και αυτό θα πρέπει να περιέχει και ένα χρονοδιάγραμμα για τις μελλοντικέ συζητήσεις και στην Ολομέλεια. Δεν έχω πρόβλημα να συνέλθουν οι σκιώδεις από την ε, Επιτροπή μας και την Επιτροπή Απασχόλησης ώστε να λύσουν το θέμα. Και όμως είμαστε στη φάση που πρέπει να έχουμε μια συμφωνία. Και αν δεν υπάρχει συμφωνία θα έχουμε δεύτερη απόρριψη. Οπότε πρέπει να είμαστε αρκετά ρεαλιστές ώστε να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Ως πρόεδρος λοιπόν, απλώς σας θυμίζω παιδιά ότι από εσά εξαρτάται το αν θα έχετε τελικά συμφωνία. Αν δεν μπορείτε, η επιλογή για την Επιτροπή και την Ολομέλεια είναι εκεί. Κύριε Ζασάντη, θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω για αυτό το θέμα. Θα χαιρόμουν αν ήσασταν ε, ε, γιατί έχουμε μόνο 15 λεπτά μετάφραση. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο έγγραφο αυτό υπάρχουν πολλά σημαντικά στοιχεία τα οποία μπορούν να επηρεάσουν ενδεχομένως την όλη κατάσταση και να μειώσουν το κόστος. Βεβαίως, ο, αν υπάρχει μία και μοναδική διαδικασία ε, η οποία θα ακολουθηθεί για την ενοποίηση, δεν θα χρειάζεται να ζητούμε εξουσιοδότηση από 27 κράτη-μέρη. Τώρα, αν αποφασίσουμε στην Επιτροπή μας να εργαστούμε την Επιτροπή Πασχόλησης, γιατί όχι. Διότι ασχολούμαστε με λεπτομέρειες πολλές φορές χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα θέματα τα κοινωνικά με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή Επασχόλης τώρα αν θα πρέπει να αποφασίσουν για τον αριθμό των φορέων που παρέχουν τις επίσης στα κράτη-μέλη θα δημιουργηθεί ενδεχομένω πρόβλημα αν κάποιος μειώσει από τρεις σε δύο τους φορές αυτούς και αν κάποιος από αυτούς ε, τους δύο εγκαταλείψει την όλη διαδικασία μπορεί να αντικαταστήθει με κάποιον άλλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις που αφορούν το έγγραφο αυτό στη δική μας επιτροπή. Βεβαίω εγώ είμαι διατεθειμένος οποιαδήποτε στιγμή <clears throat> συναντηθώ με τους συναδέλφους της Επιτροπής Πασχόλης και να καταλήξουμε στη συμφωνία. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε όλοι να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό στη δικασία. Θα πρέπει να παρακολουθήσω εκ του τι γίνεται όταν ε, συνεδριάσετε με τους ε, ε Θα πρέπει όλη αυτή η δικασία να αρχίσει αρκετά γρήγορα για να καταλήξουμε σε λύση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης σήμερα. Τώρα περνούμε αμέσω στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ όσοι δεν θα συμμετάσχουν να φύγουν. Και όπως έκαναν παλιά και ο, ε, στο, στη Βουλή των Λόρδων την εποχή των ε, βασιλέων στο παρελθόν, ζητείτε από όλους τους ανεπιθύμητους να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Παρακαλώ λοιπόν αυτό να γίνει.